Good Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω. Καθίστε παρακαλώ. Thank σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ως ήθιστε, εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, έχουμε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής μας, στο πλαίσιο αυτής της Ολομέλειας του Στρασβούργου. Δευτέρα βράδυ, ως ήθιστε έχουμε τρομερό φόρτο εργασίας. Προσπαθήστε να μπείτε ήσυχα γιατί προσπαθούμε να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ. Έχουμε μεγάλη ημερήσια διάταξη. Πρέπει να τα δούμε ένα-ένα τα θέματα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν έχουμε νομίζω πρόβλημα, εγκρίνεται το σχέδιο μέσα της διάταξης. Ανακοινώσεις για τη διερμηνία. Έχουμε όλες τις γλώσσες πριν, πλην Ιρλανδικών, Μαλτεζικών και ε, Κροατικών. Πρώτο ουσιώδες σημείο της ημερής σας διάταξης αυτής της βραδινής συνεδρίασης είναι διαρθρωμένος διάλογος με τον Αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου ζωή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχά σα καλωσορίζω. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ μαζί μα. Και μεγάλη μας τιμή που θα έχουμε την πρώτη ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, το χαρτοφυλάκιό σα. Σα ευχόμαστε καταρχά κάθε επιτυχία και πολύ τύχη για τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και βεβαίω προσβλέπουμε σε μια πολύ στενή συνεργασία στα πολύ σημαντικά ζητήματα που εμπίπτουν στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο σας, άσυλο και μετανάστευση ιδίως, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης, κοινωνικής ένταξης, που κατά τη γνώμη μας είναι εγγενές στοιχείο της προώθησης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Και βεβαίως η εσωτερική ασφάλεια για το μέλλον του Σέγγεν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του πρώτου διαθρωμένου διαλόγου που διεξάγουμε μαζί σας, θα ορίσουμε και τον ρυθμό, την τακτικότητα αυτών των διαλόγων στο μέλλον, στη διάρκεια της θητείας. Και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τις προτεραιότητες του Μαργαρίτη Σχοινά, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο που έχει αναγγελθεί. Η δουλειά επί του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει με τον ε, Επίτροπο Γιώχανσεν. Η Επίτροπος Γιώχανσεν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μαζί μας και ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει μια συνέχεια της ε, συζήτησης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, οι συντονιστέ έχουν αποφασίσει να αποστείλουν επιστολή με την οποία θα τροφοδοτούν τη διαμόρφωση αυτού του Συμφώνου Μετανάστευση και Ασύλου με τι δικέ μα σκέψει. Μετά το διάλειμμα των Χριστουγέννων, θέλουμε να επισημάνουμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε τα σχέδια της Κομισιόν σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εσωτερική Ασφάλεια της Κομισιόν, η οποία θα συζητηθεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις αρχές του νέου έτους. Ας δώσουμε πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για 15 λεπτά και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Με τον συνήθι τρόπο, συντονιστές και συνέχεια μέλη της Επιτροπής. Να σας υπενθυμίσω ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προβλέψει είναι από τις 7.30 έως τις 9 για, αυτό το πρώτο τμήμα της εμείς διάταξης. Γιατί μέχρι τις 9 θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον ε, Αντιπρόεδρο Σχοινά και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Ράιντερς για, για δικαιοσύνη και θα έχουμε και μαζί μας εκπρόσωπο της Φιλανδικής Προεδρίας, τον κύριο Τοπολάιν, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το κράτος δικαίου. Πολωνία, Ουγγαρία και Μάλτα. Αυτά θα γίνουν στο δεύτερο μισό της συνεδρίασής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Λόπες Αγγιλάρ, ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε πριν από τα Χριστούγεννα. Μια μέρα που καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ φορτωμένη για εσάς. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στις 3 Οκτωβρίου κατά την ακρόαση επιβεβαίωσής μου, το επίκεντρο της προσοχής τη συζήτηση αφορούσε βεβαίω τι προθέσει. Σήμερα έρχομαι εδώ ενώπιόν σα, για πρώτη φορά έκτοτε με τη φιλοδοξία να αρχίσουμε τη συζήτηση επί των δράσεων ή τον δρόμο που θα ανοίξουμε προς τις δράσεις. Και επαναλαμβάνω σήμερα, όπως και τότε, ότι ο τακτικός, ειλικρινής και ουσιώδης ε, διάλογος με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι ζωτική σημασίας. Αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να αναφερθώ σε τρεις κατηγορίες ζητημάτων. Μετανάστευση, άσυλο και σχετικό σύμφωνο. Δεύτερον, ασφάλεια. Και τρίτον, κοινωνική ένταξη. Και σύνδεση με το, πώς να το πω, τα θέματα που δεν αφορούν, δεν είναι αρμοδιότητα στις ΛΥΜΠΕ. Ξεκινώ από τη μετανάστευση. Γνωρίζω ότι μιλώ σε ειδήμονες και η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά στον τομέα της μετανάστευσης αλλά δεν τα έκανε όλα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι έχουμε πλέον κάνει μια σημαντική αλλαγή. Έχει υπάρξει μια μεταστροφή. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μου ανέθεσε τον συντονισμό των εργασιών για αυτό το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που είναι, ας το πούμε ειλικρινά, ο τελευταίος ελίπων κρίκος του συνολικού μοσαϊκού μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο όρος σύμφωνο είναι ένας όρος ευγενής. Γι' αυτό και πρέπει να του προσδώσουμε περιεχόμενο, όπως συμβαίνει πάντοτε με αυτούς τους ευγενείς όρους πρέπει να εξευρεθεί μια, ένα νέο είδο συνένεση για το πώς διαχειριζόμαστε και διαμορφώνουμε τις πραγματικότητες τη μετανάστευσης και πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε μέσω του συμφώνου ότι θα είμαστε σε θέση να πείσουμε τους πολίτες μας ότι η Ευρώπη μπορεί να, επιφέρει, να αποφέρει αποτελέσματα σε κάτι που διαμορφώνει και επηρεάζει τις συμπεριφορές μας, τις κοινωνίες μας, την πολιτική που ασκείται σε ολόκληρη την Ήπειρο. Για να γίνει αυτό, για να προχωρήσουμε προς το σύμφωνο δηλαδή, πρέπει πρώτα να αφουγκραστούμε. Και αυτό ξεκινήσαμε με την Επίτροπο Γιώχανσεν, ξεκινήσαμε από την Αθήνα και συνέχεια μεταβήκαμε στο Βερολίνο, στην Παρίσι, θα πάμε την επόμενη Πέμπτη στη Βουδαπέστη και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία, αν θέλετε, στις πρωτεύουσες, στη διαδικασία αυτή του αφουγκρασμού ε, των ανησυχιών που εκφράζονται. Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε από αυτές τις πρώτες επαφές προς το δρόμο για το σύμφωνο αυτό, καθώς και από τις συζητήσεις που είχαμε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων, ήταν αρκετά ενθαρρυντικά τα μηνύματα που πήρα. Έχουμε την αίσθηση ότι πλέον αναδεικνύεται μια κοινή αντίληψη, μια συναντήληψη ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποτύχουμε άλλη φορά. Η αποτυχία λοιπόν δεν είναι στο μενού και η συνολική εντύπωση που έχουμε αποκομίσει από αυτές τις πρώιμες επαφές είναι ότι υπάρχει μια σύγκληση γύρω από δύο θεμελιώδεις έννοιες. Πρώτον, ότι το σύμφωνο αυτό θα πρέπει να είναι ένα συνολικό σύμφωνο, ένα ολιστικό σύμφωνο αν θέλετε. Και δεύτερο, ότι δεν θα καταλήξουμε πουθενά αν δεν εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την ανάληψη ευθύνη. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή αυτού του συμφώνου. Μπορώ όμως να σας περιγράψω την γενική μα αντίληψη για τα βασικά στοιχεία που θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαμορφώσουν την ε, τελική μορφή αυτού του συμφώνου. Πρώτον, πρέπει να ε, υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση, λαμβανωμένου υπόψη ότι η εξωτερική και η εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης είναι αλληλένδετες και δεν μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει ξεχωριστά. Ένα νέο σύμφωνο σημαίνει ότι τα εξωτερικά σύνορα και η διαχείρισή τους θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η εσωτερική ελεύθερη κυκλοφορία που είναι εμβληματικό χαρακτηριστικό της Ένωσης μας. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται επιτάχυνση και επιχειρη επιχειρικοποίηση της Ευρωπαϊκή συνοριοφιλικής και εκτοφυλακή και η καταπολέμηση από πλευρά Ευρώπη των λαθρεμπόρων και των διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για τα κέρδη του. Επίση σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών για εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ήπειρό μα. Επίση, απαιτεί κάτι τέτοιο, η υλοποίηση διαδικασιών ασύλου, χορήγηση ασύλου, που θα είναι ισχυρές και ανθεκτικές και θα λαμβάνουν υπόψη και το ζήτημα των δευτεροβουσών μετακινήσεων. Επίση, ο πολιτικό σύνδεσμο ανάμεσα στο Σέγγεν και στο άσυλο είναι σαφή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα του συστήματο ασύλου πρώτα, για, για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Επίση, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για του νομικού δρόμου που θα ακολουθήσει η Ευρώπη ώστε η αγορά εργασίας μας να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το ταλέντο και τα προσόντα των μεταναστών βασιζόμενοι βεβαίως ε, στα επιτεύγματα που έχουμε ήδη κατακτήσει. Και τέλος χρειάζεται ε, ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης κινητοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όχι μόνο τα χρήματα και τις επενδύσεις, αλλά και το εμπόριο, τις θεωρήσεις, την κινητικότητα, τα, τις υποτροφίες Εράσμους, όλα όσα μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη ως ε, τμήμα μιας εταιρικής σχέσης αμοιβαίου ωφέλους με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Επίσης επισκεφτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα την Τουρκία, που είναι βασικός εταίρος στρατηγικής σημασίας και ζωτικής σημασίας παράγοντας σε μια ευμετάβλητη περιοχή η οποία έχει υποδεχτεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Καμία χώρα δεν μπορεί να ε, φιλοξενήσει περισσότερους ε, πρόσφυγες από ότι η Τουρκία. Επαναλάβαμε τη σημασία που έχει η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και νομίζω ότι στο σωστό χρόνο εξασφαλίσαμε ότι και τα 6 δισεκατομμύρια του μηχανισμού για τους πρόσφυγες για την Τουρκία έχουν πλέον αποδεσμευτεί. Και ας είμαστε ειλικρινεί σε ένα συνολικά ε, δύσκολο πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία να συνεχίσουν τους επαφές τους. Όπως ε, έχει επαναλάβει ε, πολλές φορές και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πάμε τώρα στην ασφάλεια στην ατζέντα για την ασφάλεια. Έχω δεσμευτεί τον περασμένο Οκτώβριο ενώπιον σα ότι θα δώσουμε προτεραιότητα και στι παραδοσιακέ και στις μοντέρνες απειλέ. Επαναδιατυπώνω αυτή τη δέσμευση του χρόνου. Θα προωθήσουμε μια νέα στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια που θα αντιμετωπίζει τομεί με ισχυρή διασυνοριακή διάσταση όπως τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, κοιμιωμένο έγκλημα, ε, συνεργασία των διοκτικών αρχών και το να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια στις, ε, στον κόσμο των πληροφοριών. Θα κοιτάξουμε και το, την εντολή της Europol. Θα ήθελα με ευκαιρία να επαναλάβω τη σημασία μια σύντομη συμφωνία για, ένα κανονισμό για να προλάβουμε την διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου online, που είναι πολύ σημαντικό για να εκριζώσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και την ε, βίαιη ε, στάση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι απειλέ ε, από το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα, λαμβάνοντα υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει τροποποιήσει τον τρόπο που λειτουργούν αυτέ οι ομάδε. Στον αγώνα κατά του κυβερνοεγκλήματο, θα προσέξουμε ιδιαίτερα την προστασία, την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών μα, ε, η σεξουαλική κατάχρηση και παρενόχληση των παιδιών online έχει αυξηθεί εκθετικά και θα δράσουμε αποφασιστικά στον τομέα αυτό. Η εξελισσόμενη φύση των απειλών στην ασφάλεια ζητούν ε, οριζόντιες προσεγγίσεις που θα ξεπερνούν το κλασικό πλαίσιο εσωτερικών υποθέσεων και τον τρόπο που νοούμε την εσωτερική ασφάλεια. Ε, και θα πρέπει το ψηφιακό, το ενεργειακό κομμάτι, της ε, χρηματοπιστωτικής υπηρεσία στην υγεία, όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και εδώ είναι η προσθέμενη αξία του χαρτοφυλακίου μου. Θα ενισχύσουμε την ε, στάση μας να προλάβουμε, να αντιμετωπίζουμε και να, αντιμε... και να εκριζώνουμε τις απειλές αυτές. Ε, τα συστήματα πληροφορικής μας θα γίνουν πιο διαδραστικά και θα αναπτύξουμε μια υγιή προσέγγιση ε, στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, ε, κατάλληλη για την ψηφιακή και παγκόσμια εποχή, με δισεκατομμύρια συνδεδεμένα αντικείμενα και συστήματα με ευαίσθητες πληροφορίες. Επομένως, είναι σημαντικό για την Ευρώπη να εξασφαλίσει ότι η κυβερνοασφάλεια και η αντοχή της των, των δικτύων πέμπτης γενιάς είναι εκεί που πρέπει. Το να προστατεύσουμε τις ψηφιακές κρίσιμες υποδομές, αυτό ε, συνδυάζεται με την προστασία φυσικά και των φυσικών υποδομών. Θα έχουμε μια ευέλικτη ε, προσέγγιση, ούτω ώστε με βάση τον κίνδυνο, ούτω ώστε να είμαστε ανθεκτικοί ε, σε όλους του κινδύνους, ε, στα drones, ε, στις, σε διάφορες απειλέ. Επαναλαμβάνω τη δέσμευση που έδωσα εδώ τον Οκτώβριο, ότι κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις μας εξορισμού θα έχει ενσωματωμένο το, το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι προσωπική δέσμευσή μου αυτή. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα είναι ένα συμπλήρωμα εκ των υστέρων ε, στη δουλειά που κάνουμε για την ασφάλεια. Θα είναι η πόρτα που ανοίγει, το κλειδί που ανοίγει τα πάντα, όλα όσα κάνουμε για την ασφάλεια. Δεν θα κάνουμε πίσω στις ε, αξίες μας, όπως θα κάνουμε πίσω και σε θέματα ασφάλειας και θα, τις προστατεύσουμε, θα τα προστατεύσουμε και τα δύο μαζί. Δέκα μέρε έχω αναλάβει τα καθηκόντά μου. Από την πρώτη μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν άρχισα να δουλεύω ε, σε αυτό το ανθρωποκεντρικό χαρτοφυλάκιο, είπα ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τις δικές σας αρμοδιότητες, τα θέματα της ΛΥΜΠΕ. Υπάρχουν και άλλοι όμως άξονες που θα πρέπει να τους δω μαζί με τους αρμόδιους επιτρόπους, ε, πέρα από αυτούς, αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα ήδη. Σας ε, ξαναλέω ότι μαζί με τη Στέλλα Κυριακίδου θα Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο ευρωπαϊκό για τον καρκίνο. Μαζί με τη Μαρία Γκάμπριελ θα έχουμε δράσεις, ούτω ώστε να καταστήσουμε μέχρι το 2025 πραγματικό τον ευρωπαϊκό χώρο ε, εκπαίδευσης. Μαζί με την Νίκολα Σμιτ θα αναδιατυπώσουμε την ατζέντα για τις δεξιότητες, ε, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ε, νέες δεξιότητες κτλ. Όλα αυτά γιατί τα κάνουμε, για να εξασφαλίσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ιστό και από αυτό να αποτελείται μια ε, συνεκτική κοινωνία του αύριο. Προστασία, ασφάλεια, δεξιότητες, κινητικότητα, ικανότητα να αντιμετωπίσουμε ένα γοργά εναλλασσόμενο περιβάλλον. Προφανώς θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών. Είναι οι νέοι Ευρωπαίοι που θα τους ε, συναπαντήσουμε τα επόμενα χρόνια και τους ε, χρωστάμε το ίδιο επίπεδο προστασίας και πρόσβασης όπως εξασφαλίζουμε στους δικούς μας πολίτες. Τους επόμενους μήνες θα αποκρισταλώσουμε όλες αυτές τις ε, δράσεις, αυτούς τους άξονες δραστηριότητας και θα εξασφαλίσω τη συμπληρωματικότητά τους με ένα κεντρικό στόχο το να οικοδομήσουμε πιο στενή, πιο αποτελεσματική, πιο ανθεκτική, πιο ισχυρή ευρωπαϊκή κοινωνία ή ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και σε κάθε φάση αυτής της πορείας ε, θα ζητήσω την συνδρομή σας. Ξεκινάω ήδη με τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα απόψε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, ε, πρόεδρε Σχοινά. Ξεκινάμε τη συζήτηση, ο συνήθως πρώτα οι συντονιστές. Κυρία Μετσόλα από το ΕΛΚ θα είναι η πρώτη. Και προτείνω να ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος με όσους ε, συναδέλφους ε, θέλουν το λόγο και τους παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι, την κάρτα, τέλος πάντων να προσελκύσετε την προσοχή της γραμματείας για να σας εγγράψουν στον καταλοκέρα Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε και στην ακροασή σα την 3η, Οκτωβρίου και σήμερα απόψε με πολλά παραδείγματα δείξατε ότι είναι ιδιαίτερα τεταμένο το χαρτοφυλόκιό σα για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου. Θα εστιάσω καταρχάς στην ασφάλεια και έχω και μια άλλη ερώτηση για την Τουρκία. Για την ασφάλεια Πώς θα ολοκληρώσουμε την Ένωση Ασφάλειας είναι το ερώτημά μου, ιδίως ό,τι αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο online. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο ποια είναι τα σχέδιά σας για την αντιμετώπιση του περιεχομένου αυτού εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία. Και στον τομέα αυτό φυσικά υπάρχουν ευαισθησίες που δεν πρέπει να τις ε, ε λησμονούμε. Εθνική δηλαδή ε, ασφάλεια και αρμοδιότητα των κρατών μελών πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, μια καλύτερη, ε, πιο γρήγορη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφόρων μεταξύ κρατών μελών και πώς ε, θα επηρεαστούν όλα αυτά από την προβλεπόμενη πλέον αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του επόμενου μήνα. Για την Τουρκία. Είπατε ότι συναντήσατε πριν από λίγε ημέρε τον πρόεδρο Ερντογάν. Είδαμε ότι όσοι ήσασταν εκεί, οι αφήξει στα ελληνικά νησιά είχαν ε, σταματήσει. Όταν φύγατε όμω, ε, άρχισαν να καταφθάνουν κατά εκατοντάδε πάλι ε, στα ελληνικά νησιά Πρόσφυγε και μετανάστες. Η προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα. πώ αντιλαμβάνεστε την κατάσταση ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ευρώπη και αν ναι, πώς πρέπει να ανταποκριθούμε ή να αντιδράσουμε. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Σίπελα από τους Ελληνικέ και δημοκράτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σχοινά που είστε εδώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρέμβασή σα. Δεν παίρνουμε και κανένα θαύμα, αλλά για να είμαι ειλικρινή, όταν μιλήσατε για την ασφάλεια και για τη μετανάστευση, δεν άκουσα και τόσες πολλές νέες ιδέες Ολιστική προσέγγιση, με τα χαρά να τη συζητήσουμε. Είναι μια προσέγγιση που ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει στην προηγούμενη θητεία, οπότε και είχαμε συζητήσει για σαφείς διαδικασίες για το άσυλο, για την νόμιμη μετανάστευση και την καλύτερη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής. Να δούμε δηλαδή ποια είναι και τα δικά του συμφέροντα, ώστε να είναι ενήμεροι καλύτερα οι πολίτες για τις ε, δυνατότητες που έχουν και γιατί τι δεν υπάρχουν. Εσεί μιλήσατε για νόμιμους διαδρόμους για, για να αντιμετωπίσουν τα συμφέροντά μας και στον τομέα της απασχόλησης. Δεν άκουσα να μιλάτε για αντίστοιχου νόμους διαδρόμους για τους χρήζοντες προστασία. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό και σε ό,τι αφορά αυτούς τους νόμους διαδρόμους για τη μετανάστευση. Αυτή η συζήτηση για την μπλε κάρτα δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχουν άλλες ιδέες για να υπερπηδηθεί το σχετικό αδιέξοδο, το σχετικό εμπόδιο στη συζήτηση. Επίσης, επιστροφές ε, πάντοτε ήταν ένα κομμάτι ε, της διαδικασίας ασύλου, είναι όμως το τελευταίο ε, στάδιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλιστεί σωστή διαδικασία. Αυτό πώς θα το εξασφαλίσετε. Ιδίω λαμβάνοντα υπόψη τι νέε ιδέε, νέε παλιέ αν θέλετε ιδέες, κάποια ανεπίσημα έγγραφα όπω είναι και από τη γερμανική κυβέρνηση που αναφέρεται σε κάποιο είδους, πώς να το πω, ε, ζώνες διέλευσης, ε, transit zones, στα εξωτερικά σύνορα. Θα ήθελα να μου πείτε ε, τι ιδέες έχετε, πώς θα οργανωθούν αυτές οι ζώνες, περί τίνος πρόκειται. Είπατε επίσης ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσε πολλές μετανάστες και πρόσφυγες σαν Τουρκία. Όχι, δεν αληθεύει αυτό. Ε, ο Λίβανος, για παράδειγμα, έχει υποδεχθεί πολλού περισσότερους μετανάστες αν συγκρίνουμε τον πληθυσμό του με τους μετανάστες και οι αφρικανικές χώρες επίσης ε, ε, φιλοξενούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από ότι η Τουρκία, άρα να μην λέμε ψέματα. Και τέλος, για την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι σημαντική για όλους τους πολίτες. Όταν μιλάμε για το κυβέρνο έγκλημα, Πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να ακούω συνέχεια ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το κυβερνοέγκλημα λόγω της ε, κακοποίησης παιδιών, της σεξουαλικής κακοποίησης, που φυσικά και είναι ένα έγκλημα, το οποίο ποτέ δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Αλλά πραγματική κακοποίηση δεν γίνεται στο διαδίκτυο, αλλά στην πραγματική ζωή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε και η διερεύνηση αυτού του φαινομένου το τελευταίο στάδιο, ε, ναι λυπούμε πρόεδρε μακρηγόρο, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στην έρευνα, στην πρόληψη αυτών των εγκληματικών πράξεων στην πραγματική ζωή και να μην χρησιμοποιούμε τέτοια παραδείγματα ω πρόσχημα ουσιαστικά για να διεισδύσουμε στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών. Ευχαριστώ. Σε περίπτωση που χρειάζεται να το υπενθυμίσω, κάθε φορά που δίνω το λόγο, να θυμάστε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 ακόμη ομιλητέ. Αν θέλετε να τα καταφέρουμε μέσα σε μια μισή ώρα, να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, α προσπαθούμε, ας προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε ευσύνοπτε, γρήγορε ερωτήσει, δύο λεπτά για του συντονιστέ, ένα λεπτό για όλου του υπόλοιπου. Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο τρόπο για να χειριστούμε την κατάσταση που έχουμε μπροστά μα. Η κυρία Ίντβολτ για τον Ρινιού. Ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπε σε αυτή την πρώτη σας παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής μας. Σύντομα, για την ασφάλεια και τη σχετική στρατηγική που ανακοινώσατε. Θα ήθελα να πω κάτι επί της ε, μεθοδολογίας. Γιατί τα τελευταία χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, η προσέγγιση ήταν ε, μάλλον ε, τσαπατσούλικη. Η Κομισιόν υπέβαλε προτάσει τη μία μετά την άλλη, χωρί να συνοδεύονται από τι αναγκαίε μελέτες επιπτώσεων και εμεί, ω Επιτροπή το ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδεχτούμε αυτό. Δεν πρόκειται να, να ξαναδεχτούμε καμία πρόταση αν δεν συνοδεύεται από μελέτη αντικτύπου. Η ε, εφαρμογή είναι αξιοθρύνητη, αξιολόγηση είναι ανύπαρκτη και όπως πολλές φορές έχουμε προβλέψει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος ε, νομικών πράξεων και συμφωνιών που έχει πιέσει για την ε, έγκριση, της, ε, έγκριση τους η Κομισιόν τελικά καταργούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα τα κάνετε καλύτερα εσεί. Δεύτερον, για τη μετανάστευση. Είπατε ότι, για, και την ασφάλεια. Είπατε για τα εξωτερικά σύνορα. Ξέρετε όμως ότι μια από τις μεγαλύτερες Πηγέ βίας στην Ήπειρο είναι η ενδοοικογενειακή βία. 2.500 έως 3.000 γυναίκες το χρόνο πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους στην Ευρώπη λόγω της ενδοοικογενειακή βίας. Εγώ δεν έχω δει ούτε διαδηλώσει ούτε και μεγάλα χρήματα για το ζήτημα αυτό. Εσείς τι θα κάνετε για το σύμφωνο μετανάστευση. Εσείς και η Επίτροπος Γιώχανσον είπατε ότι έχετε κάνει μια εκστρατεία στις πρωτεύουσε. Ναι, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθέτης. Έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε διαπραγματευτεί καλή την πίστη με το Συμβούλιο και τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το Συμβούλιο μας λέει «Α, δεν ξέρουμε τι θέλουμε ακριβώς, το κοιτάμε ακόμα» και στη συνέχεια πηγαίνετε στι πρωτα... πρωτεύουσε για να δείτε τι έχουν να σα πούνε οι άνθρωποι. Γιατί δεν έρχεστε στον νομοθέτη να σα πούμε εμεί τι θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Δεν είναι δυνατόν. Το νομοθετικό έργο το οποίο έχουμε κάνει εμεί με την υποστήριξη εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών μπορεί απλά να το πετάξετε εσεί στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχτούμε αυτό και σα το ξεκαθαρίζω προσωπικά. Είστε πλέον Επίτροπο, όχι για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου, ε, ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, αλλά για την προώθηση αυτού. Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Εμείς ε, σας έχουμε, έχουμε πει ότι είστε ο αγαπημένος μας lifestyle coach στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς θα μας προστατεύσετε από τις εσωτερικές απειλές στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δηλαδή τις αξίες μας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 των συνθήκων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι πράσινοι έχουν το λόγο. Η κυρία Στρίκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Σχοινά, γιατί είναι η πρώτη σας φορά εδώ υπό τη νέα σας ιδιότητα του Επιτρόπου. Θέλω να τονίσω ε, αυτά που είπε ε, με επιτακτικό τρόπο η κυρία Ιντβελτ, να συμμορφωθείτε με την διοργανική συμφωνία, να συνοδεύονται οι προτάσεις σας με, από μελέτη αντικτύπου όταν κρίνετε ότι θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και ταυτόχρονα να ε, δημοσιεύετε εκθέσεις με, τρόπο που θα, ε, με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπετε στα, στην ομοθέσια μας, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ελπίζω να αναλάβετε μια σχετική δέσμευση σήμερα μιας και είστε εδώ μαζί μας. Έχω ένα ερώτημα για το άσυλο. Ε, προτεραιότητα του κυρίου Σχοινά είναι, όπως μας είπε, να υπάρξει συνένεση με τα κράτη-μέλη ε, γύρω από το ζήτημα του ασύλου. Όμως εξεπλάγει ότι η πρώτη σας επίσκεψη, όχι ότι η πρώτη σας επίσκεψη ήταν στα ελληνικά νησιά, αλλά η δεύτερη επίσκεψη ήταν στην Τουρκία και όχι σε κάποια πρωτεύουσα κράτους μέλους. Ήταν ε, αρκετά μεγάλη έκπληξη. Βεβαίως, οι πρόσφυγες υπάρχουν πολλοί στην Τουρκία. Ε, όμως ο Ερντογάν ε, είναι και μια απειλή για τους πρόσφυγες γιατί τους χρησιμοποιεί ως ε, ε, όπλο. Έχει απειλήσει μάλιστα να απελάσει στο, στην πράσινη ζώνη που έχει δημιουργηθεί στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας 1,5 εκατομμύριο ε, πρόσφυγε. Γι' αυτό και έχω συγκεκριμένα ερωτήματα να σα θέσω. Εσεί τι ακριβώς ε, συμφωνήσατε με τον Ερντογάν. Θεωρείτε ότι αυτή η buffer zone είναι ε, περιοχή ασφαλή όπου μπορούν να επιστραφούν οι Σύριοι πρόσφυγες. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ο Ερντογάν δεν θα στείλει Σύριου πρόσφυγε στη βορειοανατολική ε, Συρία. Και ποιε θα είναι οι επιπτώσει για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις και πώς ακριβώς θα παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Ταρντίνο. Κύριε Ταρντίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Επίτροπο, πρόσφατα πήγατε στην Τουρκία μαζί με την Επίτροπο Γιώχανσεν και τονίσατε ότι η επίσκεψη αυτή ήταν μια ευκαιρία για να δείξατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Τουρκία στρατηγικό εταίρο με τον οποίο συνεργάζεται εν ώψη του γεγονότος ότι έχει και το στάτους της υποψήφιας χώρας. Είναι η νιωστή φορά που η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό του Ερντογάν, ο οποίος ζητάει απλώς λεφτά από τα, από τα κονδύλια των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως η συμφωνία με την Τουρκία έχει να κάνει με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στην πραγματικότητα η Τουρκία αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά της. Εσείς πήγατε όμως να την διαβεβαιώσετε ότι οι κρουνοί χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα σταματήσουν. Δεν σας φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση ε, και αυτό το κράτος δεν σέβεται το στυλ ε, και τον τρόπο ευρωπαϊκής ζωής. Επίσης, την επόμενη άνοιξη θα παρουσιάσετε το πακέτο για τη μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει για το, στο θέμα του Δουβλίνου. Τι θα κάνετε μέχρι την Άνοιξη. Είσαστε σε θέση να παρουσιάσετε μία πρόταση που θα λύσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν, δεν μας είπατε τίποτα. Επίσης, με ποια λεφτά, με ποιο προϋπολογισμό θα φτιάξετε μία πλειοψηφία για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάνει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για τα χρήματα τα οποία δίνεται σε ΜΚΟ ε, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ε, Μεσόγειο. Οι προηγούμενοι επίτροποι δεν δώσαν απάντηση. Εσείς μπορείτε να δώσετε απάντηση σε αυτό το θέμα. Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά που δίνονται σε ΜΚΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέω κύριος Προκατσίνη. Κύριε Σχοινά. Καλή δουλειά καλή τύχη πάνω απ' όλα. Είσαστε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο οποίος μου γεννά τις μεγαλύτερες ελπίδες. Για λόγους ουσίας, όχι για τυπικούς λόγους. Γιατί στην πραγματικότητα λίγα μας δώσατε, αντικαταστήσατε μία λέξη με μία άλλη στον τίτλο του χαρτοφυλακίου σας. Και ενώ μιλούσατε για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, ε, επειδή ορισμένοι θεωρούσαν ότι αυτό ήταν πολύ επιθετικό, ε, μιλιταριστικό, φασιστικό, εσείς τους ακούσατε και αλλάξατε αυτή τη λέξη. Λες και η κουλτούρα μας, οι αξίες μας, ε, αν, αν τις προστατεύουμε, σημαίνει ότι επιτιθέμεθα σε κάποιου άλλου. Εμένα μου φαίνεται παλαβό αυτό, αλλά τέλο πάντων. Τέλος πάντων, τώρα δεν μιλάτε πια για προστασία, αλλά για πρόθεση. Μια και αλλάξατε αυτή τη λέξη. Σε τι θα αλλάξει η δράση σας. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί η στήριξη απέναντί σα από κάποιες κοινοβουλευτικέ ομάδες σας δίδεται, σα σας δόθηκε μάλλον μόνο και μόνο γιατί αλλάξατε αυτό το όνομα. Μένει λοιπόν μια αμφιβολία για τις αρμοδιότητές σα κυρίως σε ό,τι αφορά τα θέματα μετανάστευση. Δεν κατάλαβα ποια είναι η γραμμή οριοθέτηση. Ε, ανάμεσα στα δικά σας καθήκοντα και στα καθήκοντα της Επιτρόπου Γιώχανσον για τα θέματα της μετανάστευσης. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η νόμιμη μετανάστευση και η ασφαλής μετανάστευση είναι το πρώτο θύμα από την λάθρο μετανάστευση, από την παράνομη μετανάστευση. Επίσης, θα αντιμετωπίσετε την παράνομη ε, μετανάστευση και κυρίως μιλάω εδώ για τους οικονομικούς μετανάστες, που είναι ένα ακαθόδες θέμα. Τέλος, για το θέμα της Τουρκίας. Δεν θέλω κι εγώ να σας γυρνάω το μαχαίρι στην πληγή. Νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη στην Τουρκία ήταν ένα μήνυμα υποταγής απέναντι σε έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι αξιόπιστος και είναι επιθετικός. Γκουε. Η Κορνιλιά Ένστ. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Σχοινά, θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Είπατε ότι θέλετε με την κυρία Γιώχανσεν να αναλάβετε τον συντονισμό του μηχανισμού ασύλου και μετανάστευση. Μα τι σημαίνει αυτό. Τι θέλετε ακριβώς να συντονίσετε δηλαδή. Εννοείται με τον συντονισμό, με, την, με τον όρο συντονισμό να πηγαίνετε από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη και να παρακαλάτε την Ουγγαρία αν μπορεί η Βουδαπέστη να πάρει άλλου τρει ε, πρόσφυγες. Πώς ακριβώς το φαντάζεστε και ποια ακριβώ θα είναι η στάση σα απέναντι σε εμά. Εμεί, στην προηγούμενη θητεία με, δύο, με πλειοψηφία δύο τρίτων υποβάλαμε μια πρόταση για προοδευτική υποδοχή προσφύγων από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Τι θα γίνει με αυτή την πρόταση. Θα την λάβετε υπόψη, θα βασιστείτε σε αυτήν ή έχετε σκοπό να, να μας φέρετε μια τελείως καινούργια πρόταση. Ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στη δική μας δουλειά. Επίσης, το δικαίωμα ασύλου, το ατομικό δικαίωμα ασύλου σας αφορά, είναι κάτι που το λαμβάνετε υπόψη σας, με βάση την, την ε, συνθήκη της Γενέβης ή απλά ε, επειδή ε, επικεντρωθήκατε μόνο στο ζήτημα των επιστροφών. Επίσης, είπατε για αξιολόγηση, για διασυνοριακό κίνδυνο, εγκληματικότητα κτλ αυτό θα το αξιολογήσετε και όσον αφορά τους πρόσφυγες στα εξωτερικά σύνορα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στα κροατοβοσνιακά ε, σύνορα επικρατεί μια κατάσταση κολαστηρίου. Τους παίρνουν τα λεφτά, τους παίρνουν τα κινητά, κυνηγούν ανθρώπους μέσα σε ποτάμια. Αυτέ, αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα σας απασχολήσουν ή όχι. Τρίτον, έχετε σκοπό να αξιολογήσετε τα χρηματοδοτικά κονδύλια που δίνετε στην Τουρκία ότι κατευθύνονται πραγματικά και καταλήγουν εκεί για, για, για, για, για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Έχετε ε, κάποια συγκεκριμένη εικόνα. Και τέλος, δεν είπατε τίποτα για το resettlement, για την επανεγκατάσταση, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Ποια, ποια μορφή θα έχει αυτή η επανεγκατάσταση. Ε, Παρακαλώ, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Θα πρότεινα τώρα να πάμε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 Κυρία Αντιπρόεδρε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την πρώτη έτσι διευρυμένη συζήτηση στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Πράγματι, σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία. Είναι μεγάλο το χαρτοφυλάκιο, είναι πολλές οι ευθύνες. Θα επικεντρωθώ στο ένα λεπτό σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, ακούστηκε μια συγκεκριμενη ερωτηση ακουστηκε μια κριτικη που σας ασκήθηκε για την επίσκεψή σας στην Τουρκία προσωπικά εγώ πιστεύω ότι ήταν αναγκαία η επίσκεψή σας στην τουρκία και σε ό,τι αφορά την άποψή μου θα σας το ζητούσαμε γιατί όταν ζητούμε από την τουρκία μια συνεργασία αποτελεσματική ειδικά στο θέμα το μεταναστευτικό θα πρέπει να συζητήσουμε και μαζί τους. εδώ όμως έρχομαι να σας ρωτήσω ευθέως τι πρόκειται να γίνει με τη συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας με το δεδομένο κύριε αντιπρόεδρε ότι αναμφίβολα από πλευράς του Προέδρου Ερντογάν δεν τηρείται πλέον η συμφωνία. Και όχι μόνο δεν τηρείται, αλλά με τρόπο εξαιρετικά προκλητικό επισημαίνεται ότι ε, μπορεί κατά το δοκούν να εκβιάζει με τη συμπεριφορά προς αυτήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα, σας παρακαλώ, ένα λεπτό καθένα. καθένας. Ο Ευχαριστώ πολύ τηλεγραφικά κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, Αντιπρόεδρε που είστε εδώ και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να αλλάξει η νοοτροπία που υπάρχει σε ορισμένε χώρε και σε ορισμένου συμπολίτε μα για τη μετανάστευση. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Οι μετανάστε δεν είναι απειλή, δεν είναι πρόβλημα, είναι ε, μία ανάγκη, είναι και μια ευκαιρία και η Κομισιόν μέχρι στιγμής έχει εστιάσει ε, στο, στην πιο αρνητική πλευρά, την καταναγκαστική πλευρά, δηλαδή την επιστροφή ε, και τις αποθήσεις ενδεχομένως στην Τι θα γίνει όμως με τη νόμιμη μετανάστευση, τι οδηγίες έχουμε και την κυκλική μετανάστευση, την ένταξη των μεταναστών. Και υπάρχει μια ιδέα για ένα ευρωπαϊκό ταμείο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση άμεση τοπικές αρχές, δηλαδή δήμαρχοι ε, των πόλεων. Τι έχετε να μας πείτε πάνω αυτό και το τελευταίο για τα ασυνόδευτα παιδιά, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Δύο σύντομες ερωτήσεις ο κύριος Τουντοράτσε για τη μετανάστευση. Σε αυτό το ε, συμφωνώ. Ε, πρέπει να εξορροπήσετε την ευθύνη για αλληλεγγύη από τη μία και εξωτερικά όταν θα πάτε σε τρίτες χώρες να δεχθούν ε, τους επιστρεφόμενους, αν θέλετε, μέσω των νόμων διαδρόμων να τις πείσετε στις χώρες αυτές. Τι γίνεται με αυτές τις χώρες και τα κράτη-μέλη Πώ θα τα πείστε να κάνουν περισσότερα από ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πιλωτικά προγράμματα αναφέρατε. Δεν έχουν ε, κάνει τίποτα στην πράξη, ενώ συμβολικά μπορεί να δίνουν μια καλή εικόνα, αλλά ε, είναι ελάχιστε οι θέση, 20-30 και το 5 5G. Ποιο θα αναλάβει αυτό που έγινε ε, το έργο King, του Julian King. Το 5G λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μήπως έφυγε το τρένο από το σταθμό σε σχέση με το τι έχουν οι ήδη ορισμένα κράτη-μέλη. Κυρία Κάνκο, ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ Επίτροπε και ιδίως που τονίσατε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα πρόσφατα Είχατε, όπω είπατε, επικοδομητικό γύρο συνομιλιών ε, στην Άγκερα με την Τουρκία. Η Τουρκία φυσικά ε, και φιλοξενεί του περισσότερου πρόσφυγες στον κόσμο. Έχουμε κάποια στοιχεία από το 2018 από την ύπατη αρμοστία ε, για του πρόσφυγε. και γι' αυτό θέλω να πω στην κυρία Ζήπελα από του Ασυλιστέ ότι δεν συμφωνώ μαζί τη γιατί τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πράγματι η Τουρκία φιλοξενεί του περισσότερου πρόσφυγες στον κόσμο. Και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για την τον έλεγχο της συγκράτησης μετανάστευσης ζητείτε ε, μετά από την επιστροφή σας ε, η ε, Τουρκία να συνεργαστεί γιατί είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος και υποψήφιος αλλά για κάποια ο Ερντογάν έχει μιλήσει με αρνητικά λόγια. Είναι ρεαλιστικά όλα αυτά πριν από λίγες εβδομάδες έλεγε ότι θα ανοίξει τις πύλες για να πλημμυρίσει με πρόσφυγες και μετανάστες την Ευρώπη εάν δεν συνεχίζα, μάλλον δεν κάναμε αυτό που ήθελε σε ό,τι αφορά τη Συρία. Τι θα γίνει λοιπόν και με αυτό το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο είναι πολύ ρευστά τα όσα γίνονται σε εξωτερικά σύνορα. Πώς θα το λάβουμε αυτό υπόψη και για την Τουρκία. Μια χώρα σαν την Τουρκία μπορεί ποτέ να είναι αυτή η χώρα μέλος της Ένωσης. Κύριε Σχοινά, για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και των ευρωπαϊκών αξιών θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η αλληλεγγύη, ασφάλεια ή αξιοπιστία είναι κάτι που η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι είναι σημαντικές αρχές για εμάς. Όταν θα διαπραγματεύεστε με αυτή τη χώρα λοιπόν να το έχετε και αυτό υπόψη. Ένα λεπτό. Εάν δεν μιλάτε ε, για ένα λεπτό, έχουμε πρόβλημα. Ο καθένας να σέβεται το ένα λεπτό. Ε, κύριε Ρέσλερ, κύριε Σχοινά, έχετε ένα πολύ πλατή χαρτοφυλάκιο. Θέλω να εστιάσω στη μετανάστευση. Και παρότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, πολύ πλατή, πολύ μεγάλο, πρέπει να δούμε και τις νόμιμες οδούς, ε, τα βιώσιμα ε, τι βιώσιμες μεταναστευτικέ ροές, συνεργασία με τις χώρε που βρίσκονται καθοδόν και συνεργασία με τις χώρε που παράγουν μετανάστευση. Και να δούμε και τις βασικές αιτίες μετανάστευσης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρέ μεταναστευτικέ πιέσει. Το ερώτημά μου είναι να μας εξηγήσετε λιγάκι τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για να υποστηρίξετε τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα και πώς αναγνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μεταναστευτικές οδούς. Η κυρία Γκυγιόμ, ένα λεπτό. Εάν μας προτείνετε ένα νέο σύμφωνο, είναι γιατί τα προηγούμενα πακέτα, σχέδια κτλ. απέτυχαν. Και αν απέτυχαν, είναι γιατί μπλοκαρίστηκαν στον τριμερή διάλογο και αυτό γιατί. Γιατί πολλά από τα κράτη-μέρη μπλόκαραν αυτά τα κείμενα. Και γιατί, να συνεχίσω το γιατί, γιατί μερικοί δεν θέλουν τους μετανάστες. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι έχετε πραγματικά την πρόθεση να αποσύρετε το κείμενο για το Δουβλίνο, ε, το κείμενο αυτό για τις διαδικασίες, να το αντικαταστήσετε με κάτι άλλο, αυτό που σημαίνει ότι μόνο η θέση των κρατών θα περάσει και όχι του Κοινοβουλίου και θα ε, το αντικαταστήσετε με ένα σύστημα ε, κατανομής από τα εξωτερικά σύνορα. Και αν απαντήσετε καταφατικά, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην εμπειρία κάποιων κρατών μελών, όπου θεωρούν, θεωρούμε ότι οι μετανάστες δεν πρέπει να μπουν στην επικρατειά μας, βρίσκονται σε χώρες αναμονής, σε κέντρα κλειστά και επειδή δεν μπαίνουν δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν έχουν δικαιώματα για το άσυλο και είναι απλώς το μόνο που, τους, ε, που μπορεί να του πέσει το κεφάλι με μια απόφαση απέλαση. Άμα το επιβεβαιώσετε, τότε μιλάμε για γενικευμένη κράτηση σε κλειστά κέντρα. Αυτό ε, νομικός πώς, εθικός, πώ με βάση τους ε, κανόνες του διεθνού δικαίου, είναι σωστό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει. Τα ευρωπαϊκά κείμενα για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ασύλου έχουν φοβερές ε, διαφορές τον τρόπο που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί μιλάμε το κάθε κρατό μέλο ότι έχει τις δικές του, ε, τα δικά του δικαι... προνόμια και δικαιώματα. Θα κάνετε κάποια επικαιροποίηση για, αυτό το, για αυτή τη δουλειά. Μιλήσατε επίσης ε, για τη σημασία με τις τρίτες χώρες, τις χώρε προέλευση, τι χώρες εταίρου. Τι κάνετε από κοινού με τον είπα το εκπρόσωπο, ε, τον κύριο Μπορέλ, για αυτό το θέμα. Κύριε Μπράιερ, πράσινη. Επίτροπε, άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε για την στρατηγική ασφάλειας που θα μας προτείνετε. Και ανησυχώ, λόγω των παρελθουσών ε, εμπειριών που ήταν μια στρατηγική επιτήρησης, όχι ασφάλειας πάντα λέτε ότι για να αλλάξουμε μια νομοθεσία λέμε ας πούμε ότι η παλιά νομοθεσία δεν ήταν ικανοποιητική, έγιναν εγκλήματα κτλ. Ε, Όμω, ε, αν έχουμε ένα κράτο, α πούμε, αστυνόμου, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι θα είμαστε πιο ασφαλεί. Προσοχή λοιπόν όταν προτείνετε το νέο κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά επανάληψη, ακύρωσε την νομοθεσία για να κατο, καταγράφουμε ε, ιδιωτικέ συνομιλίε όταν δεν υπάρχουν υποψίε και να φυλάσσουμε αυτά τα δεδομένα. Έχετε καμιά πρόθεση, ε, Επίτροπε, να κάνετε νέα ε, πρόταση για τη φύλαξη δεδομένων. Ε, μια και κάνετε πρόσφατη επίσκεψη στην Τουρκία. Ποια είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσεων για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ Europol και Τουρκίας. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέιλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απογοητεύτηκα λίγο από την έλλειψη λεπτομεριών των εισηγητικών σας παρατηρήσεων και λίγο με ανησύχησε το η στάση σας απέναντι στην Τουρκία. Το ότι είπατε ότι κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα από την Τουρκία όσον αφορά τους πρόσφυγες, εκτός αν εννοούσατε βεβαίως ε, εννοούσατε ότι η Τουρκία έχει συμβάλει στη δημιουργία προσφύγων. Και μετά είπατε ότι θα εξασφαλίσετε και ενισχυμένο ρόλο για την Ευρωπόλ. Και εδώ θέλω να πω, στην τελευταία σας επίσκεψη στην Τουρκία, ε, συζητήσατε το θέμα τη ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με την Τουρκία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμεί ω Κοινοβούλιο έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τον ορισμό του εγκλήματο, τη τρομοκρατία. Δεν υπάρχει δήλωση επιπτώσεων και ακούμε ότι οι διαπραγματεύσει βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά δεν έχουμε λάβει καμία λεπτομέρεια, λεπτομερή πληροφορία σε σχέση με αυτό. Όσον αφορά την ε, online παραπληροφόρηση, ε, η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ε, είναι ένα ε, θέμα ε, το οποίο βεβαίως ε, αντιτίθεται σε εκείνους που έχουν τους κυρίαρχους αν θέλετε. Πού όμως ακριβώς μπαίνει η γραμμή ανάμεσα στην προστασία από την παραπληροφόρηση και την λογοκρισία. Ο κύριος Ζήκατς για την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο που η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές κάπως προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Ε, όποιος έχει παρακολουθήσει τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα έχει καταλάβει ότι μέσω του διαδικτύου ε, πραγματοποιείται διανομή και εμπορία υλικού παιδικής πορνογραφίας. Από αυτή την άποψη η Ευρωπόλ ασκεί εξαιρετικά τα καθήκοντά της και εκτελεί ένα, επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο. Πώς θα υποστηρίξετε την Ευρωπόλ στο μέλλον, στα καθήκοντά τη αυτά. Ρουίς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά και τον Αντιπρόεδρο Σχοινά για τι εξηγήσεις που μα έδωσε μέχρι τώρα. Θα συμφωνήσω με όσα υπόθηκαν για τις δυνατότητες ε, ε, που προσφέρουν οι μετανάστες ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και με όσα είπε ο συνάδελφος Χαβιέρ Μωρέ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για αυτή ε, την νέα προσέγγιση για το μεταναστευτικό σύμφωνο. Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, ξέρουμε ότι η αποτυχία είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το δεχθούμε. Πώς να θα αποφύγουμε την αποτυχία. Τελικά είναι ε, ένας ε, τρόπος αυτός ε, το να έχουμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή του Συμβουλίου αφήνοντας και καταλείποντας το επίπεδο φιλοδοξίας που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν ποια νέα δυναμική θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι δυνατή μετά από το γύρο συνομιλιών σας με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Μάρκετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να σας πω ότι την πέμπτη τελευταία εβδομάδα από το γερμανικό Spiegel σε ένα βίντεο αποδεικνύεται, τουλάχιστον ε, υπάρχουν στιγμιότυπες σε αυτό το βίντεο, ότι γίνονται αποθήσεις στον Εύρο και ε, Επομένω, υπάρχουν ε, αποδείξεις που δείχνουν ότι όσο δεν δίνει απαντήσει η Κομισιόν ε, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ε, εσείς τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά και το κράτος δικαίω Κομισιόν. Και το δεύτερο, όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά δεν είναι και τόσο καλή. Ε, και μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι εικόνες ντροπή αυτά που βλέπουμε. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Σαλάχ που έχει δημιουργήσει μια οργάνωση, οι οποίοι μας δίνουν ελπίδες, αλλά μετά αυτούς τους ανθρώπους φυλακίζουμε. Ε, και ο συγκεκριμένος καταγορήθηκε και ορισμένα πράγματα τα οποία φυσικά δεν μπόρεσαν να αποδειχθούν. Ε, θέλω να σας ρωτήσω τι κάνετε με αυτές τις περιπτώσεις. Μήπως τελικά βοηθάμε τους διακινητές αντί να βοηθάμε τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν κάτι για να λυθεί το πρόβλημα εκεί. Εσείς ένα λεπτό κύριε Μπαρέν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σχοινά που ήρθατε εδώ. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι κάποια κράτη όπως η Ισπανία για παράδειγμα πρόσφατα πέρασαν νομοθεσία για το ε, επιγραμμικό περιεχόμενο που μας ανησυχεί. Φαντάζομαι ότι θα πείτε ότι είναι νωρί για να το κρίνουμε. Εγώ όμω θέλω να σα ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σα για τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά την τυχή τη ασφάλεια και την νομοθεσία περί επιγραμμικού περιεχομένου. Τι προτίθεστε να κάνετε για να είναι το διαδίκτυο πιο ασφαλές, αν αυτό βέβαια είναι δυνατόν. Είναι απαρχαιωμένες κάποιες διατάξεις ε, ε, και τι θα γίνει με την ελευθερία έκφρασης και ανταλλαγές πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σεβαστό. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Σχοινά, σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις που μας δώσατε σήμερα. Ένα από αυτά που είπατε και που το χαιρετίζω είναι η εστίαση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, στην ε, στρατηγική για την ασφάλεια και σημείωσα επίσης ότι έχετε κάνει μια εκστρατεία με την Επίτροπο Γιώχανσεν σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε, όπου είμαι βέβαιος ότι πρέπει να είχατε πολύ σημαντικές συζητήσεις με τους ομολόγους σας. Όμως, κάτι που χάνεται όταν δεν πηγαίνετε σε μικρότερα μέρη και όχι πρωτεύουσε, είναι οι καθημερινές εμπειρίες ε, που ζουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, όπως η μαμά ε, που γνώρισα στον παιδικό σταθμό του παιδιού μου, ε, που μου έλεγε ότι μέρα μεσημέρι της κλέψαν το αυτοκίνητο, άνθρωποι από ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος και το ερώτημά μου είναι ε, εσείς τι με καλείτε να της πω αυτής της γυναίκας όταν με ρωτήσει την επόμενη φορά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά μου. Ευχαριστώ. Κύριε Σχοινά, για το ζήτημα της μετανάστευσης ε, μιλήσατε για τους διακινητές και το οργανωμένο έγκλημα. Πώς μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να υποστηρίξει την, ε, τον αγώνα εναντίον των διακινητών στην Κεντρική Μεσόγειο. Θα ξαναρχίσετε τις ε, επιχειρήσεις. Δεύτερο, για την ασφάλεια. Μιλήσατε για την ενέργεια, τις μεταφορές και την υγεία ως ε, προστιθέμενη αξία της ασφάλειας. Συμφωνώ. Όμως τι, τι, ποια είναι η στάση σας απέναντι στη διεθνή διαφθορά. Η διεθνής διαφορά επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των πολιτών μας. Μην, ξεχνάτε λοιπόν και τον σύνδεσμο με τις οργανώσεις του ε, οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά την ασφάλεια. Οπότε, εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Μαγκίτ. Κύριε Σχοινά, σε καμία, άλλη, ε, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μειώνονται οι αντισλαμικές, ισλαμοφοβικές ε, επιθέσεις παντού βλέπουμε ενίσχυση ε, αυτών των φαινομένων. Όταν διάβασα τις προθέσεις σας, με εξέπληξε το γεγονό ότι ενώ μιλάτε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και συμφωνώ απολύτω, δεν αναφέρεστε καθόλου στην καταπολέμηση τη Ισλαμοφοβία. Θεωρώ ότι η, η, η θέση σα μπορεί να συμβάλλει στην ε, εξάλληψη της ε, σύνδεσης του εγκλήματος της τρομοκρατίας με, το, με, τον, με την Ισλαμοφοβία. Εσείς λοιπόν, επειδή εγώ μπορεί να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται, ε, τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να μην ε, μένει κανείς πίσω σε αυτήν την Ευρώπη. Ο κύριος Μπουσαδέ. Ευχαριστώ να μιλήσω στα ισπανικά σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρέμβασή σας. Σας συγχαίρω και για τον ορισμό σας. Σύντομα, ο σύντροφος μίλησε για Ισλαμοφοβία. Εγώ ήθελα να σας θέσω ένα πρόβλημα και ε, πλήττει αυτό ε, τον τρόπο ζωής. Είναι οι χριστιανοί οι οποίοι διώκονται και σε αυτούς θέλω να αναφερθώ. Ε, σε χριστιανικές κοινότητες αντιμετωπίζουμε επίσης προβλήματα και επίσης μια ΜΚΟ που μεταφέρει ε, μετανάστες από τη Λιβύη στην Ευρώπη. Ο Πενάν σε μένα tweet έλεγε αρχίζουμε την αποστολή μας 72, φτάνουμε στην άλλη άκρη της ε, ακτής, της όχθης τι θα γίνει από την Κομισιόν ε, για τη δράση αυτή των ΜΚΟ και ποιος τελικά θα υπερασπιστεί τον Ευρωπαϊκό Τρόπο. Θα ε, βοηθήσετε τα κράτη και για τις ε, πολιτικές γονιμότητας στην Ευρώπη. Γιατί τελικά σε κάποια χρόνια δεν θα είναι κανένας που θα μπορεί να υπερασπιστεί τον Ευρωπαϊκό Τρόπο ζωής. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πήγα στη χώρα σας, στην Ελλάδα, λέει ο Μποσελάγκε. πήγα στα hot spot και είδα και εγώ την κατάσταση Φαίνεται ότι χιλιάδες άνθρωποι παγώνουν, ε, ε, κοιμώνται έξω, δεν έχουν ε, φάρμακα, πολύ στοιχειώδεις συνθήκες, τους λείπουν τα βασικά. Ούτε από την Επίτροπο Γιώχανσεν που τη ρώτησα το ίδιο, δεν να την απάντηση. Θα προσπαθήσετε να υπάρξει εκένωση ιδίω των ε, ανσυνόδευτων και των πιο ευπαθών ε, από τα κράτη αυτά με την ε, συνεννόηση με τα άλλα κράτη-μέλη. 1.200 είναι αυτά τα συνόδευτα παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι επίση που ζουν υπό αναξιοπρεπεί συνθήκε και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι. Εσεί θα τη δώσετε τη μάχη αυτού του ανθρώπου που υποφέρουν τόσο καιρό. Μπαρτόλο. Μπαρτόλο. Ο τελευταίο ομιλητή ήταν αυτό και δεν νομίζω ότι ξέχασε κανέναν ο τελευταίος ομιλητής. Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή αξιολόγησε τις συνέπειε τη δημογραφική ύφεση τη Ευρώπη και τι μα περιμένει μέχρι το 2050. Είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί όταν μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση και νόμιμες μεταναστευτικές οδούς, ε, μιλάμε αποκλειστικά για ε, εργατικά χέρια με δεξιότητες. Δεν χρειαζόμαστε και άλλου είδους εργαζόμενους στην Ευρώπη όμως. Και δεδομένου ότι στη συζήτηση έγινε αναφορά ε, σε ένα διαβόητο non-paper, δεν πιστεύετε ότι αυτά τα χαρτιά τα οποία κυκλοφορούν ε, πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα μιλάνε για επαναπατρισμό, έτσι. Μόνο για επαναπατρισμό κάνουν λόγο αυτά τα διαβόητα χαρτιά που κυκλοφορούν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μίλησαν όλοι όσοι ήθελαν να πάρουν το λόγο. Έθεσαν τα ερωτήματά τους και τις ανησυχίες τους προς τον Αντιπρόεδρο κύριο Σχοινά. Κύριε Σχοινά, έχουμε ακόμα μισή ώρα πριν από το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, γιατί είναι πολύ βαριά η σημερινή ατζέντα. Έχουμε τον Επίτροπο Ράιντερς και την ε, Υπουργό του Πινάιρ για την Ουγγαρία, Πολωνία και τη Μάλτα. Πολύ βαρύ και αυτό το σημείο. Κύριε Σχοινά, κάντε το καλύτερο, το καταδύναμη. Έστω και μία λέξη για κάθε ερώτημα, αν αφιερώσετε, ε, θα νομίζω θα μας ε, ικανοποιήσετε. Το χειρότερο είναι να αγνοήσετε κάποιους από αυτούς που ε, εξέφρασαν τις ε, απόψεις τους. Κάντε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε να απαντήσετε τώρα όσο μπορείτε και αν θέλετε μπορείτε τα σημεία τα οποία δεν καλύψατε τώρα, μέσα αυτή τη μισή ώρα που μας μένει, να τα απαντήσετε γραπτός, αργότερα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους και σας Πρόεδρε και τους ομιλητές, τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Ε, σε προηγούμενες ζωές ε, πάντα παρατηρούσα εκ του σύνεγγυς ε, ως παρατηρητής τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είχα τους λόγους μου. Τα περισσότερα από τα θέματα που συζητούνταν εδώ, αργά ή γρήγορα γινόταν θέματα τα οποία απασχολούσαν τις υπηρεσίες στις οποίες εργαζόμουν εγώ. Γι' αυτό λοιπόν Χαιρετίζω τον ενθουσιασμό, τη ζωτικότητα, την ζωντανή συζήτηση με την οποία και τον τρόπο με τον οποίο συνομιλείτε εσείς. Ε, πάντα έτσι συνομιλείτε ε, και θίγεται μια πλατιά, ε, ένα πλατή φάσμα θεμάτων. Να ξεκινήσω από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τις πολλές ερωτήσεις που υποβάλατε και που αφορούν με κάποιο τρόπο αυτό το θέμα, αυτή την έννοια και αυτό το χαρτοφυλάκιο, το οποίο όπως ξέρετε είναι νέο, δεν υπήρχε πριν σε αυτή τη μορφή. Αντίθετα από τις απόπειρες πολλών να θεωρήσουν ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ένας οδοστρωτήρας που υπάρχει μόνο και μόνο για να συνθλίψει οτιδήποτε βρίσκει στο δρόμο του ή αντίθετα από την αντίληψη άλλων που θεωρούν ότι είναι ένα δίπολο. Είμαστε ένα δίπολο. Εμείς και οι άλλοι. Εμείς και οι βάρβαροι. Ε, εγώ θέλω να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι έτσι τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Για μένα ο ευρωπαϊκός τρόπο ζωής, και το είπα αυτό στην ακρόαση, είχα την ευκαιρία να το εξηγήσω, ήταν κάτι που έμοιαζε με καθρέφτη. Που από... εκφράζει αυτό που είναι η Ευρώπη σήμερα. Το τι είμαστε, το με τι μοιάζουμε, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Είμαστε τώρα λιγότερο από το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είμαστε περίπου το 20% όμως του παγκόσμιου πλούτου και ξοδεύουμε το 50% των κοινωνικών δαπανών παγκοσμίως. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε μια χαρά είναι αυτό. Είναι ένα μοντέλο ζωή που μα και κοινωνία που μα αρέσει. Ή μπορούμε να θέσουμε σοβαρά ερωτήματα για το πώ μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα επιτεύγματα σύν το χρόνο. Πώ θα μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την επιτυχία που είναι η Ευρώπη, η σημερινή Ευρώπη, στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Εγώ ποτέ δεν θεωρούσα ότι αυτό σημαίνει αποκλεισμό, μίσος. Εγώ πάντα το εννοούσα και το κατανοούσα ως προσπάθεια ένταξης. Η προστασία και η προώθηση έχει κάποια, κάποιες αποχρώσεις. Το καταλαβαίνω. Ζούμε σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ε, το κοινοβούλιο ζήτησε να το λάβει υπόψη. Η πρόεδρος αυτό το έλαβε υπόψη. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι ε, θεωρούν ότι ο όρος προστασία ενέχει κάτι το επιθετικό. Είναι σαν να θέλουμε να προστατεύσουμε κάτι δικό μας αποκλείοντας κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ε, βάλαμε την πρόθεση που είναι κάτι πιο θετικό χωρίς αποκλεισμούς. Κάνα πρόβλημα. Εγώ έχω αγοράσει πολλά βιβλία στη ζωή μου αλλά ποτέ δεν αγόρασα ε, ένα βιβλίο λόγω του τίτλου στην πρώτη σελίδα. Πάντα λόγω του συγγραφέα ή λόγω του περιεχομένου αγόρασα εγώ τα βιβλία μου. Και περιμένω ότι ο κόσμος θα κρίνει αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, με βάση το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου και ε, τον συγγραφέα και όχι τον τίτλο του χαρτοφυλακίου. Αυτό το θέμα έχει να κάνει και με πολλά άλλα σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις σχέσεις μου με διάφορους άλλους επιτρόπους, κυρίως την Επίτροπο Γιώχανσον, αλλά και με άλλους. Να επαναλάβω αυτό που είπα και στην ακρόαση, ότι με βάση την επιστολή για την αποστολή μου, έχω συγκεκριμένα καθήκοντα και θέλω να μεγιστοποιήσω και να βελτιστοποιήσω τη δουλειά των επιτρόπων που δουλεύουν στη δική μου ομάδα. Δεν σημαίνει ότι θα τους υποκαταστήσω. Όχι, δεν σκοπεύω, δεν έχω τη φιλοδοξία να αντικαταστήσω κανένα επίτροπο, αλλά έχω κάθε προσδοκία και εσείς την έχετε να κάνουμε ακριβώς αυτά που υποσχεθήκαμε να κάνουμε. Ε, μισθοανάστευση, ασφάλεια, ε, το σύμφωνο, ευρωπαϊκός χώρος ε, εκπαίδευσης, ε, ευρωπαϊκές δεξιότητες, όλα αυτά θα πρέπει να τα προωθήσω μαζί με τους επιτρόπους, όχι εν απουσία τους. Τώρα, επανέρχομαι σε πολλά από αυτά που θέσατε. Ε, κράτησα λεπτομερείς σημειώσεις και ελπίζω να μην με προδώσουν. Να ξεκινήσω με την ασφάλεια καταρχήν. Είπα ξεκάθαρα νομίζω ότι η μελλοντική στατική ασφάλειας θα είναι μια ασφάλεια που θα αντιμετωπίζει. Τα πάντα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογική πρόοδο, αλλά και τις παραδοσιακές απειλέ, τεχνολογικές και νέες απειλέ δηλαδή, αλλά και παραδοσιακές απειλέ. Θα ήταν σφάλμα να δώσουμε έμφαση ε, στον ένα άξονα ει βάρος του άλλου. Δεν μπορούμε να έχουμε ψηφιακέ υποδομές εάν δεν έχουμε ε, σοβαρή απόκριση για τι απειλέ που έχουμε στη ε, φυσικέ υποδομέ μα. Δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνοαποκρίσεις εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές στα πυρηνικά μας εργοστάσια, στα λιμάνια μας, ε, στις φυσικές μας υποδομές. Αυτά πάνε μαζί. Η έμφαση ε, στις διασυνοριακές απειλές είναι προφανής. Γιατί εκεί έχουμε την ισχυρότερη νομική βάση. Εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μαζί με, το, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Εκεί μπορούμε να δικαιολογήσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, σέβομαι απολύτως τα θέματα όπως αυτό που αναφέρθηκε από τη Σόφη Ιντβελτ για την ε, οικιακή βία. Θα συνεργαστώ με την ε, Επίτροπο Γιούροβα και τον Επίτροπο Reinders για μια νέα στρατηγική για το φύλλο που την έχει ανακοινώσει η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν ήδη και είναι προφανές ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτό το πλαίσιο. Το ίδιο αφορά και τον τομέα της βίας κατά διαφορών θυμάτων, ε, ευάλωτων πληθυσμών και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να σας ε, επισημάνω ότι δεν πρέπει να διαφοροποιούμε το φυσικό επίπεδο σε αντιδιαστολή με το ψηφιακό. Και τα δύο μαζί. Είτε το ένα είτε το άλλο και τα δύο είναι το ίδιο και τα διασυνδέουμε αυτά σε ένα νέο έγγραφο στρατηγικής που στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο τώρα. Για την ασφάλεια και πάλι. Δεν συμμερίζομαι το φόβο πως ε, ασφάλεια σημαίνει επιτήρηση. Καταλαβαίνω ότι ε, υπάρχουν αυτοί οι φόβοι, αλλά νομίζω ήμουν σαφής όταν είπα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα τα ε, ε χρησιμοποιήσουμε ε, ως πρόσχημα για την ε, προτάσεις μας. Είπα ότι είναι ένα, εξ, είναι ένα εμπροστοβάρες, όχι εξπόστ. Θα γίνει κάτι το οποίο προηγείται. Και έχουμε νομίζω τα εχέγγυα ως προς αυτό. Έρχομαι στην Τουρκία που ενδιαφέρει πολλούς και πολλές από εσάς από διάφορες πτυχές κατανοητά όλα θεμητά όσα είπατε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν αποφασίσαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να πάμε στην Τουρκία. Δεν είπαμε για να φτιάξουμε βαλίτσα και να πάμε στην Τουρκία. Αφού είμαστε στην Αθήνα, περάσουμε απέναντι και να πάμε στην Τουρκία. Όχι, δεν έγινε έτσι. Είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις με τους Υπουργούς Εσωτερικών ε, στο επίσημο γεύμα του Συμβουλίου, όπου ε, βολιδοσκοπήσαμε τις απόψεις των Υπουργών ε, για το κατά πόσο η τέτοια επίσκεψη θα ήταν χρήσιμη και υπήρχε, θα έλεγα περιέργως, σχεδόν ομοφωνία από τα κράτη-μέλη ότι είναι μια επίσκεψη που θα είναι χρήσιμη για την Ευρώπη. Τώρα, παρά το αυτό. Δεν πήγαμε χωρίς να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει κατανοητή ο λόγος της επισκεψής μας από ε, την Τουρκία. Η πρόεδρος Φοντρελάιν συνομίλησε μακρόν με τον πρόεδρο Ερντογάν πρώτης επισκέψεώς μας όπου ε, κατέστη σαφές, απολύτως σαφές το πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη. Δεν πήγαμε εκεί για να ξεκαθαρίσουμε και να λύσουμε όλο το φάσμα ε, των ε, ευρωπαϊκών, ε, τουρκο-ευρωπαϊκών σχέσεων που δεν και στην καλύτερη στιγμή, ούτε για να λύσουμε το πρόβλημα της Συρίας ή άλλα προβλήματα, αλλά για να μεταφέρουμε τρία πολύ απλά μηνύματα, τα οποία εδώ μπορώ να σας τα επαναλάβω. Πρώτον είπαμε, γεια σας, είμαστε η νέα ομάδα. Μπορεί να φαίνεται ε, λιγότερο σημαντικό από ότι είναι. Αλλά δεν ήταν τόσο σταθερές οι σχέσεις με, και οι επαφές με την προηγούμενη ομάδα, άρα ήταν σαφές ε, ότι θέλαμε να μας δουν ως νέους συνομιλητές. Δεύτερον, ε, κυρία Ζήπελ, τους ευχαριστήσαμε διότι ναι πράγματι είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο. Ίσως όχι κατά κεφαλήν, πάντως σε νούμερα είναι με βάση την είπατε αρμοστή για τους πρόσφυγες και τα στοιχεία της και τους ευχαριστήσαμε διότι θεωρούμε ότι καταβάλουν μια προσπάθεια. Ναι, με τη δική μας την υποστήριξη όμως παρόλα αυτά φιλοξενούν 4 εκατομμύρια απεγνωσμένες ψυχές που σημαίνει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει ε, να τους ευχαριστήσουμε, να τους το αναγνωρίσουμε τέλος πάντων. Και το τρίτο, τους είπαμε, ακούστε θα συνεχίσουμε να ε, ενεργούμε για τη μετανάστευση, η ιστορία, η πραγματικότητα και το παρελθόν μας καταδικάζουν αν θέλετε στο να το κάνουμε. Και κυρία Μητσόλα, ναι, είναι αλήθεια. Όσο ήμασταν εκεί, πράγματι ήταν μηδενικέ οι αφήξει στα ελληνικά νησιά και όταν φύγαμε ξανάρχισαν ε, να φεύγουν τα σκάφη. Αλλά Ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε ε, σε αυτό ακριβώς το ίδιο πλαίσιο για τη διαχείριση μετανάστευσης μάλλον δεν ήταν συζήτηση για γεωπολιτικά θέματα, για δεδομένα ή για τα μείζωνα ζητήματα, τη διεύρυνση και τα λοιπά, τις εξορρυκτικέ δραστηριότητε. Αυτά είναι ξεχωριστά ζητήματα και τα εξετάζουμε σε διαφορετικό πλαίσιο. Θεωρούμε όμω ότι αυτή η επίσκεψη ήταν σημαντική, ήταν αναγκαία και συνολικά νομίζω άφησε κάποιε προπτικές ανοιχτέ. Δεν συμφωνήσαμε με την Τουρκία ε, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ε, τα κονδύλια που δίνουμε για ε, τους πρόσφυγες. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτά να πηγαίνουν απευθεία στο κράτος και αυτή τη μέθοδο εμείς όπως ξέρετε δεν τη δεχόμαστε και προτιμούμε να χρηματοδοτούμε ε, τους φορείς του ΟΗΕ, της ΜΚΟ και κατευθείαν τις τοπικές κοινότητες επιστρέφουμε τα έξοδα της υγειονομικής περίθαψης όχι εκ των προτέρων όμως αλλά ε, τα τιμολόγια πρώτα πρέπει να παραλάβουμε και εν συνεχεία καταβάλουμε τα ποσά. Σε ό,τι αφορά την χρησιμότητα ε, του κατά πόσον θα πρέπει μετά ε, να ενεργούμε, έχουμε και το ποσό τώρα το οποίο δεσμεύτηκε, 6 δισεκατομμύρια, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την συνεργασία με την Τουρκία. Θα ήταν λάθος. Και έρχομαι στο σύμφωνο. Ποιο είναι το σημείο Ένα επιχείρημα δεν το για πρώτη φορά. Το έχω συζητήσει νομίζω διεξοδικά μαζί σας και στη διάρκεια της ακρόασης. Σε καμία περίπτωση αυτή η νέα αφετηρία, αυτή η νέα αρχή δεν θα παραγνωρίσει ή θα βάλει στην άκρη το πολύτιμο έργο του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι εάν Υπήρξε κάποια πρόοδο στην προηγούμενη προσπάθεια. Αυτή η πρόοδο ακριβώ είναι χάρη σε εσά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν ερχόμαστε εδώ για να σα ακούμε σαν σχολιαστέ, σαν παρατηρητέ, αλλά ω ε, νομοθέτε, ε, εσεί δηλαδή είστε νομοθέτε, διότι το έργο σα, το επιτυχημένο έργο σα, ε, είναι εδώ και δεν θα χαθεί. Αλλά αντίθετα θα μας βοηθήσει. Δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, άρα θα διαφυλάξουμε αυτό το έργο. Η αφετηρία όμως πρέπει ξεκάθαρα να είναι αυτά τα δύο θεμελιώδη κείμενα, από των οποίων δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Δεν φταίτε εσείς, παραλαμβάνω, το γνωρίζω, το αντιλαμβάνομαι. Η Ένωση συνολικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μεταρρύθμιση των διαδικασιών του Δουβλίνου. Θα πρέπει λοιπόν να είναι στο επίκεντρο αυτό αυτής της νέας αρχής που θα κάνουμε μαζί με τα πολλά άλλα θέματα τα οποία ανέφερα. Θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε ένα πακέτο με πράγματα που έχουν νόημα για όλους. Γιατί πρέπει να χτίσουμε συνένεση και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα κοινά συμφέροντα γύρω από το σύμφωνο που ε, θα παρεμποδίσει κάποια κράτη-μέλη να το ξεχαρβαλώσουν. Επομένω, θα πρέπει να το φτιάξουμε και να το διασφαλίσουμε αυτό το σύμφωνο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιδέε που έχουν υποβληθεί γραπτώς και το Κοινοβούλιο θα υποβάλει τέτοιε ιδέες. Είναι πάντα ευπρόσδεκτες και είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή που χρειαζόμαστε αυτό το βασικό υλικό για να χτίσουμε το τελικό οικοδόμημα. Εσείς βλέπετε πολλά έγγραφα να κυκλοφορούν από πολλές διαφορετικές χώρες, αλλά τίποτα δεν θα πρέπει να σας κάνει να πιστέψετε ότι κάποιο από τα κείμενα είναι η τελική απόφαση, είναι το τελικό κείμενο. Όχι, τελική ε, ευθύνη, το τελικό κείμενο θα το ετοιμάσει η Κομισιόν. Λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη για συνένεση, για μια προσέγγιση ευεργετική για όλου, αλλά και την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Δεν θα υποβάλουμε κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε συμφωνία, το οποίο όμω θα είναι μη λειτουργικό στην πράξη. Και, να το πάω και λίγο παραπέρα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υποβάλουμε τίποτα εάν δεν ακούσουμε πρώτα, αν δεν μιλήσουμε σε όλους και δεν εντοπίσουμε πρώτα ε, που θα προσγειωθεί αυτό το σύμφωνο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει δύο φορές πάνω σε αυτό το θέμα. Μία αποτυχία θα ήταν τρομακτική επιτυχία για την Ευρώπη που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουμε αυτό το ρίσκο να το αναλάβουμε. Θα εξατλήσουμε λοιπόν κάθε περιθώριο καλής θέληση συνεισφορών, ιδεών, ούτως ώστε να τα φτιάξουμε τα πράγματα σωστά. Να το πάω και ακόμα πιο μακριά και να σας πω ότι έχουμε την αίσθηση από αυτόν τον αρχικό γύρο επαφών με κυβερνήσεις και από τους βουλευτές εδώ ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Ε, υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα θετική. Ε, φυσικά η πολιτική περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι λίγο διαφορετική. Είναι ένα νέος κύκλος, μια νέα αρχή, όλοι κάνουν προσπάθεια για να δείξουν το καλό τους πρόσωπο. Ε, έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε ορισμένα κράτη-μέλη που είναι θετικά για μια συμφωνία, θα συνεισφέρουν προς μια συμφωνία και ελπίζουμε ότι όταν έρθουμε ενώπιόν σας κάπου την ε, άνοιξη του 2020 να σας υποβάλουμε κάτι που θα έχει νόημα. Να επισέλθω και σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν. Πρώτον για το Brexit. Είναι ξεκάθαρο ότι η ασφάλεια θα αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν όσον αφορά τη μελλοντική σχέση που θα σμιλέψουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ασφάλεια θα είναι το, ζωτικό ελάχιστο, αν θέλετε, οποιασδήποτε μελλοντική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας τα μάτια στραμμένα στην περίοδο μετά το Brexit. Ταυτόχρονα βέβαια δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα και δεν θα είναι μέλος του χώρου Σέγγεν. Από αυτή την άποψη είναι προφανές ότι το βάθος των σχέσεων δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο το βάθος που απολαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στρατηγικό σε σε στρατηγικά ζητήματα και κατά τη μεταβατική περίοδο θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Τώρα, όσον αφορά την Κροατία, με ρωτήσατε. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτές τις κατηγορίες κακοποίησης που έχουν αποδοθεί και χειριζόμαστε τέτοιου είδους κατηγορίες με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Όσον αφορά την, ε, Κροατία, τη, για τις κατηγορίες χρήσης βίας από συνοροφύλακες θα πρέπει να συζητηθούν και να διερευνηθούν. Με σοβαρό τρόπο και με πιστικό τρόπο. Βρισκόμαστε σε στενές επαφές με τις κροατικές αρχές και η Επίτροπος Γιόν Χάνσεν με ενημέρωσε χθες ότι συζήτησε το θέμα αυτό εκτενώς με τον ε, αρμόδιο Κροάτι Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει αυτές τις κατηγορίες κακοποίησης. Είναι λοιπόν ένα θέμα που το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό. Για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είπα στη διάρκεια της ακροασής μου και επαναλαμβάνω και σήμερα ότι για μας οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αποτελούν τμήμα της λύσης. Δεν είναι το πρόβλημα. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επιτελούν ε, αξιοσέβαστο έργο στην Μεσόγειο θα πρέπει να προστατεύονται αλλά οι δράσεις τους θα πρέπει να εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση των καταστάσεων αυτών να είναι πιστική και αποτελεσματική. Είχαμε τη συμφωνία για τον εντοπισμό και την διάσωση, αυτή τη μίνι συμφωνία στη Μάλτα τον Οκτώβριο με ορισμένα κράτη-μέλη. Δυστυχώς δεν έτυχε συμφωνία ευρύτερη στο Συμβούλιο. Ενδεχομένως γιατί τα κράτη-μέλη περιμένουν και το σύμφωνο για τη συνολική λύση. Όμως όσον αφορά την, τον εντοπισμό και τη διάσωση στη Μεσόγειο και τις μη κυβερνητικέ οργανώσει χρειαζόμαστε μια διαρθρωμένη, μια δομημένη λύση και όχι ε, λύσεις ad hoc που είδαμε στο παρελθόν και που δυστυχώς δεν απένιμαν δικαιοσύνη. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχω πει επανειλημμένος ότι η κατάσταση που επικρατεί στα νησιά δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Έχω πει προσωπικά ότι η Μόρια με πληγώνει ως Ευρωπαίο και ως Έλληνα. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι η Ελλάδα εκ μέρους της Ευρώπης είναι μόνη της όσον αφορά τη διαχείριση μιας πρωτόγνωρης μεταναστευτικής ροής η οποία χωρίς συστημική βελτίωση μέσω δίκαιου επιμερισμού βαρών και ενισχυμένη αλληλεγγύη, δεν μπορεί ποτέ να ανταποκριθεί και να προσφέρει τις κατάλληλες ε, λύσεις. Εμείς από το Στρασβούργο και τις Βρεξέλλε μπορούμε να κάνουμε διάφορες διαγνώσει, όμως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να τους προσφέρουμε ε, όλη την αλληλεγγύη που χρειάζονται, όχι μόνο χρηματοδοτικά κονδύλια και ad hoc ε, ε, κανόνες και βοήθεια, αλλά και μέσω της μεταρρύθμισης το, της νομοθεσίας για το άσυλο και τη μετανάστευση. Διότι χωρίς μια τέτοια μεταρρύθμιση η Ελλάδα και οι άλλες χώρες πρώτης εισόδου δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταφέρουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη. Εγώ ελπίζω ότι η Ευρώπη θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα όσον αφορά την κοινωνική ένταξη τα επόμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα διότι πιστεύω ότι βαθμιαία οι κοινωνίες μας συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για αναγκαιότητα, πρόκειται για προτεραιότητα. Δεύτερον, διότι τι οι νέοι Ευρωπαίοι οι ίδιοι θα μας ζητήσουν τα δικαιώματα που τους χρωστάμε. Τρίτον, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα καλύπτει υπό τη νέα μας πρόταση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλήσιο, πλέον και τη μακροπρόθεσμη κοινωνική ένταξη. Άρα θα έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για να, ζητώ, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με αυτά που είχαμε από τα Ταμεία Μετανάστευση που αφορούσαν ε, την βραχυπρόθεσμη ένταξη, οπότε είμαι πολύ αισιόδοξο. Έχω και άλλα τέσσερα λεπτά λοιπόν στη διάθεσή μου, οπότε θέλω να σας πω για την, Ισλαμο... για την Ισλαμοφοβία και τον αντισημετισμό και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το ζήτημα αυτό. Ίσως δεν το γνωρίζετε γιατί έγινε μετά την ακρόαση, όμως σε μια τελευταία διόρθωση του χαρτοφυλακίου μας, μου, μεταφέρθηκε το, το χαρτοφυλάκιο ε, της ισότητας στην κυρία Γιούροβα και το, η αρμοδιότητα για τον διαθρησκευτικό διάλογο και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού ανήκει πλέον σε μένα, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Για μένα ο αντισημιτισμός, η Ισλαμοφοβία και οτιδήποτε σχετίζεται με τη ρητορική μίσου είναι πλέον ασυ... είναι πλήρω ασύμβατο με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Θα το αντιστρέψω μάλιστα το επιχείρημα και θα πω ότι αυτό που μα καθορίζει είναι ακριβώ το γεγονό ότι είμαστε σε θέση να είμαστε κοινωνίε όπου αυτές οι ιδεολογίες είναι απαράδεκτες. Συμφωνώ ότι υπάρχει ενισχυόμενος κίνδυνος όσον αφορά τον αντισημιτισμό και την Ισλαμοφοβία. Δεν θα, σας, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό μαζί σας και σας διαβεβαιώ ότι θα κινητοποιήσω όλα τα όπλα στη φαρέτρα μου. Θα έχουμε ε, συνεχή και τακτικό διάλογο με τις κοινότητες αυτές αλλά και με τη δική σας Επιτροπή, ώστε με θετικό τρόπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα ζητήματα αυτά. Κύριε Σχοινά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι προσπάθειε σα. Βεβαίω θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερο, Μάλλον εκτιμάμε ιδιαίτερο το γεγονό ότι αξιοποιήσατε το χρόνο σας. Άλλα 30 δευτερόλεπτα από την κυρία Ζίπελ και μετά άλλα 30 δευτερόλεπτα στον Επίτροπο. Γιατί υπάρχει ένα, ένα ε, συμπληρωματικό σχόλιο από την κυρία Ζίπελ, αλλά όχι πάνω από 30 δευτερόλεπτα, κυρία Ζίπελ. Ναι, με μπερδεύουν με την κυρία Ζίπελ διαρκώ. Η κυρία Ιντφελτ, λοιπόν. Ναι, ο κύριος, ο πρόεδρο ε, διορθώνει. Ευχαριστώ πολύ για τις... Ε, ε, εκτενή σα απαντήσει. Μία μικρή παρατήρηση για κάτι που είπατε στην αρχή σχετικά με την ενδοκαιγενική βία που οδηγεί σε 3.000 θανάτους το χρόνο στην Ευρώπη και δεν είναι καθόλου αμεληταίο το ζήτημα αυτό. Είπατε ότι θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό μέσω της στρατηγικής για την ισότητα. Όχι, όχι. Δεν είναι ζήτημα ισότητας. Είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Όταν υπάρχουν 3.000 θάνατοι κάθε χρόνο εξαιτία της βίας που ασκείται εναντίον τους, πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και όχι ζήτημα ισότητας των φύλων. Point taken. Μάλιστα. Το σημειώνουμε. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω ότι στις αρχές του 2020 θα δούμε ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Europol και τουλάχιστον 8 χωρών Αφρικής και Μέσης Ανατολής και συμπεριλαμβανής της Τουρκίας. Περιμένουμε πληροφορίες από, την Κομισιόν, περιμένουμε εγκαίρως αυτές τις πληροφορίες. Δεύτερον, καλύπτουμε. Καλούμε τον Αντιπρόεδρο Σχοινά τέλη Ιανουαρίου ξανά για να μας ενημερώσει για το γύρο που κάνετε στα ε, ευρωπαϊκά κράτη, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μαζί με την Επίτροπο Γιώχανσον. Ε, οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να στείλουν μία επιστολή στην Επιτροπή εν, ε, δεδομένου του ότι περιμένουμε το σύμφωνο Ασύλου και μετανάστευση. τον Ιανουάριο. Θα το συζητήσουμε λοιπόν αυτό. Φαντάζομαι θα έχουμε χρόνο να ξαναδούμε το θέμα των νόμιμων οδών μετανάστευση. που είναι τόσο σημαντικό και το έθιξαν πολλοί βουλευτές σε πολλέ από τις ερωτήσεις τους. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, για τι νόμιμες οδού μετανάστευση. τι προσφέρει, ποιε είναι αυτέ ε, στο τελευταίο σχέδιο του πακέτου ασύλου και μετανάστευσης. Και τώρα έχουμε την Επίτροπο του Πουράινεν, ε, Φιλανδή υπουργό και τον Επίτροπο Ρέιντερς. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Σχοινά που χρησιμοποίησε όλο το διαθέσιμο χρόνο για να μας απαντήσει. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και κυρίως καλά Χριστούγεννα, αν τον ξαναδούμε πριν το τέλος του χρόνου so much. Now, please stay in the room. Μην βγείτε από την αίθουσα. Μην υποτακτήσετε, γιατί Still one hour and a half and three important... έχουμε ακόμα μια μισή ώρα και τρία σημαντικά θέματα. We're Τρία επόμενα σημεία θα πρέπει να τα συζητήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ουγγαρία, Πολωνία και Μάλτα είναι τα τρία επόμενα σημεία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 Συνάδελφοι. Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό. Είναι έκτακτη αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ε, γίνεται την ίδια στιγμή με την Ολομέλεια. Τι να σας κάνω όμως. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε τρία σημαντικά σημεία. Καταρχάς έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις With... με την Προεδρία του Συμβουλίου που εκπροσωπείται από την ε, Υπουργό του Πουράινεν. Καλώς ήρθατε στη Λίμπε. Και θα ακούσουμε σημαντικά σημεία Καταρχάς, τα συμπεράσματα της ε, Προεδρίας ε, του Νοεμβρίου του 2019 για την αξιολόγηση του ετήσιου διαλόγου για το κράτος δικαίου. Δεύτερον, η συνέχεια που θα δοθεί στην πρόταση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Γνωρίζουμε ότι επί Φιλανδικής Προεδρίας μια δεύτερη ακρόαση στα πλαίσια του άρθρου, άρθρου 7.1 σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία οργανώθηκε ε, στο ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η Φιλανδική Προεδρία προσκάλεσε το Κοινοβούλιο να παραστεί σε ένα άτυπο πρωινό. Μας κάλεσε να παραστούμε. Πριν δηλαδή ε, συγκληθεί το Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών. Η κυρία Ντελβό Κόρφιντ και η κυρία Ίντφελτ ήταν πρόεδρος, που είναι πρόεδρος τη ομάδα παρακολούθηση για το κράτο δικαίου εκπροσώπησαν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην άτυπη αυτή συγκέντρωση, συνάντηση. Θέλω να επαναλάβω ότι λυπούμεθα για το γεγονός ότι παρότι ζητήσαμε να προσκληθούμε στην ίδια τη συνεδρίαση, μας καλέσατε απλώς αυτή την άτυπη συνάντηση για να παρουσιάσουμε τη θέση μας στο Συμβούλιο. Σε ένα άτυπο πλαίσιο. Επομένως, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας. Καλωσορίζω παρόλα αυτά την κυρία Τίτη του Πουράινεν, Υπουργό Εσωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη ΛΥΜΠΕ, που θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της Προεδρίας και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Με συνεχεία θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Επίτροπο Ράιντερς, Υπουργό για θέματα δικαιοσύνης. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν για αυτό το σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Και τέλος, οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σύντομες ερωτήσεις. Σύντομες. Γιατί. Γιατί έχουμε μόνο μια μισή ώρα συνολικά για να ολοκληρώσουμε αυτά τα σημεία. Το σημείο για την Ουγγαρία, το επόμενο σημείο με τους δύο ίδιους ομιλητές για την Πολωνία και τέλος θα έχουμε λίγα λεπτά για να ακούσουμε κάποια πράγματα, την παρουσίαση των συμπερασμάτων δηλαδή. Ε, μετά την αποστολή στη Μάλτα της Επιτροπής Λίμπε, που έγινε εκτάκτος και επιγόντος πριν από καμιά εβδομάδα, μέσα στο Δεκέμβριο δηλαδή. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς την Υπουργό του Πουλάινεν για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, αγαπητοί βουλευτές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Βλέπω πολλούς φίλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ, για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την κοινή συζήτηση για το κράτος δικαίου. Με μεγάλη μου χαρά έρχομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας. Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως ξέρετε, ήταν βασική προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Προσωπικά ε, εργάστηκα εργοδό πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα ως πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Για πολλού λόγους. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκέ αξίε. Αντιμετωπίζουμε όλο και πιο δύσκολε συνθήκε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι προσδοκίες των πολιτών μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και περισσότερες. Και εν μέσω όλων αυτών δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω απ' όλα μια κοινότητα αξιών. Το κράτος δικαίου είναι στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ακρογωνίας λήθος όλων των δράσεών μας. Παράλληλα, έχει και μια πρακτική λειτουργία. Το κράτος δικαίου οι ελλείψεις μάλλον του κράτους δικαίου επηρεάζουν όλα τα στρώματα ε, κοινωνίας, ε, την Ένωση, το κράτος, ε, τις τοπικές αρχές, τις εταιρείε και βεβαίως τελευταίους τους πολίτες. Ας πάμε στο σημερινό μας θέμα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ καταρχά στο διάλογο για το κράτο δικαίου που γίνεται στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζήτησε το θέμα τη ενίσχυση του σεβασμού του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το συζήτησε τρει φορέ τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Η εστίαση των συζητήσεων ε, ήταν για την ενίσχυση των εργαλείων του κράτους δικαίου της Ένωσης και της δημιουργίας ε, συνέργειας μεταξύ αυτών των εργαλείων. Η βασική λέξη, λέξη κλειδί είναι η πρόληψη. Εστιάσαμε στο να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποτρέψουμε πολύ νωρί τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός μας στόχος ήταν ο διάλογος ε, στο, Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρός, πιο ουσιαστικός για το κράτος δικαίου. Μετά την πρώτη συζήτηση στο Σεπτέμβριο, στείλαμε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη για το πώς θα γίνει ο διάλογο αυτό μια γενική συζήτηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα υπόψη ε, και τι θετικέ και τι αρνητικέ τάσει. Προτείναμε επίση ε, η νέα ετήσια έκθεση ε, της Κομισιόν για το κράτος δικαίου να χρησιμοποιείται ως ε, πλαίσιο για αυτό το διάλογο στις γραπτές απαντήσεις και στη συζήτηση τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών ήταν έτοιμες να προχωρήσουν όπως προτείναμε εμείς. Δηλαδή, φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα της Προεδρίας ε, και τα υποστήριξαν 26 κράτη-μέλη. Αυτά τα συμπεράσματα είναι μια καλή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και τη δημιουργία συνεργειών με τον κύκλο για το κράτο δικαίου που έχει δημιουργήσει η Κομισιόν. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα, θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική πρόληψη των προβλημάτων με επικοδομητική συζήτηση και συνεργασία. Φίλοι μου, θα ήθελα να πάω τώρα στο άρθρο 7.1 και την σχετική διαδικασία στο διαφορά την Ουγγαρία. Όπως ξέρετε, οργανώσαμε μια πρώτη ακρόαση για την Ουγγαρία το Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που λάβαμε την αιτιολογημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου. Θεωρήσαμε ότι είχε φτάσει η στιγμή για να κάνουμε την πρώτη ακρόαση. Αυτή η ακρόαση ήταν μια γενική ακρόαση με όλα τα θέματα που, και αυτά που συμπεριλάμβανε η πρόταση του Κοινοβουλίου. Καταρχάς έδωσε στην Ουγγαρία την ευκαιρία να μιλήσει, να, ακούς, να παρουσιάσει τις απόψεις της. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η δεύτερη ακρόαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου. Σε αυτή την ακρόαση επικεντρωθήκαμε σε τρία θέματα. Ελευθερία έκφρασης, ακαδημαϊκή ελευθερία και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά τα θέματα είναι τα πιο προβληματικά. Αυτά εντοπίστηκαν από τις περισσότερες αντιπροσωπείες στην πρώτη ακρόαση. Και στις δύο ακροάσεις τα άλλα κράτη-μέλη έδωσαν την ευκαιρία, μάλλον χρησιμοποίησαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στην Ουγγαρία και με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι οι ακροάσεις αυτές έγιναν μέσα σε επικοδομητικό πνεύμα, ε, ειλικρινή συζήτηση, αλλά με σεβασμό. Στο τέλος της ακρόασης η Προεδρία ε, ετοίμασε διαδικαστικά συμπεράσματα ότι δηλαδή το Συμβούλιο θα παραμείνει αρμόδιο για το θέμα αυτό. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς γι' αυτό το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να ενημερώνεται για τις απόψει του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό, στην αρχή της πρώτης ακρόασης, ε, σε επαφέ που είχαμε το Κοινοβούλιο, ενημερώθηκα για τις απόψει του Κοινοβουλίου και συναντήθηκα με τον Λόπεθ για να προετοιμαστώ και με την κυρία Ντελβό Σκόρφιλ μαζί με την ε, Κροατία και τη Γερμανία που είναι οι άλλες προεδρίες του τρίου. Και στην περασμένη, στην ακρόαση ε, της περασμένης εβδομάδας ετοίμασα, οργάνωσα ένα άτυπο πρόγευμα με προσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και χάρη σε αυτό το πρόγευμα κάναμε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία που αφορά την Ουγγαρία. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή τώρα Λίμπε για την καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό και γεμάτο προκλήσεις θέμα, φίλοι μας. Η διασφάλιση και η ενίσχυση των κοινών μα αξιών είναι κρίσιμο καθήκον. Απαιτεί κοινέ προσπάθειε όλων των θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών. Θα ήθελα να συνεργαστούμε προ αυτό το σημαντικό στόχο και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ του Πουράνη, εκ μέρους της Λαδικής Προεδρίας που λύγει. Όμως τώρα ας αρχίσει η συζήτηση. Προτείνω να ακούσουμε καταρχάς ε, την κυρία Ντελπο Κόρφιλτ, ε, την εισηγητριά μας και έπειτα οι Σκιώδης θα πάρουν το λόγο. 1,5 λεπτό ο καθένας θα πρότεινα και μετά ένα λεπτό υπόλοιποι που τους καταγράφουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και καμιά δυο κάμερες που μαγνητοσκοπούν. NTV 24 και TV Polsat που μας ζήτησαν να βιντεοσκοπήσουν live ε, τις εργασίες μας και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, τους το επιτρέπουμε. Οπότε προχωράμε στη συζήτηση. Βλέπω να σηκώνονται κάρτες. Παρακαλώ τηρήστε το χρονογόρευση γιατί έχουμε και την Πολωνία και έχουμε και τη Μάλτα. Ξεκινάμε με την εισηγήτρια. Λοιπόν, Κορφίλ, τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία, λέει η ομιλήτρια για τη συνεργασία που είχαμε. Η Προεδρία είχε επαφή και ενημέρωνε το Κοινοβούλιο, όπως είπε ο Λόπεθ Αγγιλάρ, η πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και η επίσημη παρουσίαση έκθεσης ε, του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, κάτι το οποίο ακόμη το περιμένουμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και που είναι εδώ σήμερα και ε, στο ε, γεύμα εργασία που αναφέρθηκε. Πρέπει να υπάρχει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, μια ειλικρινή σχέση εργασίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και έχετε και εσείς κάθε συμφέρον το κάνετε, γιατί τη δική μας την εμπειρία, η τεχνογνωσία που είναι μακροχρόνια για την Ουγγαρία μπορείτε να την αξιοποιήσετε και δεν είναι στα δικά μου χέρια απλά, αλλά πολλοί άλλοι είναι έμπειροι εδώ στο Κοινοβούλιο. Εδώ και δέκα χρόνια και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αυτό το άτυπο πρόβλημα που είχαμε πριν από την ακρόαση δεν είναι και το πιο ικανοποιητικό ως ε, τρόπο συνεργασία, αλλά τέλο πάντων ήταν θετική η συνεργασία μα σε αυτό το πρόβλημα και όλα τα κράτη-μέλη ήταν παρόντα, πολλοί υπουργοί ήταν παρόντε και Χάρη στο στένος και την εργασία της Φινατικής Προεδρίας ελήφθη δέσμευση από τα κράτη-μέλη. Ήταν ενήμερα για την κατάσταση, ήξεραν περί τίνος πρόκειται και πολλά κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν σε αυτό το πρόβλημα ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για αυτό το φάκελο και δεν θα το εγκαταλείψουν. Και από τους δύο επιτρόπους άκουσα ότι είναι προσιλωμένοι στο θέμα και θα συνεχίσουν να εργάζονται από αυτού. Ακολούθησε ακρόαση. Και κλεισμένο των θυρών υποτίθεται ότι θα γινόταν. Δεν μας είχαν προσκαλέσει. Θέλω να πω ότι αυτό είναι σοβαρό. Ε, εκείνο το πρωί υπήρξε ένα tweet ε, live από τον πρόσωπο της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Ε, συνεχώς και μάλιστα με προσβολές και δυσφημιστικά σχόλια Νομίζω ότι είναι μια, ίσως η πρώτη από τις πρώτες φορές που κάτι τέτοιο συμβαίνει και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Με τη Φιλανδική Προεδρία ε, ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί έκτοτε. Προσπαθούμε να το επικαιροποιήσουμε το φάκελ και εσείς και εμείς, σαν την εξαρτησία της δικαιοσύνης, ε, καθημερινή ελευθερία. Εδώ έχουμε όχι απλά όχι βελτίωση, αλλά και επιδείνωση κατάσταση. Στο πρόγευμα τα είπαμε διαμακρών. Όμω, έχουμε και ένα νέο στάδιο. Σήμερα έχουμε και την πολιτιστική διάσταση. Στρέφεται κατά του πολιτισμού η Ουγγρική κυβέρνηση. Περιορίζει όλες τις πτυχές της ελευθερίας Και περνάμε μία πάρα πολύ ανησυχητική διαχωριστική γραμμή, κόκκινη γραμμή που εκεί μπορούν να, να ανακαλούν, ε, να πάβουν διευθυντές καλλιτεχνικούς, να αποφασίζουν τι έργο θα παιχτεί κτλ. Τώρα περιμένουμε τι θα γίνει με την Κροατική και την Γερμανική Προεδρία. Ελπίζουμε να δείξουν το ίδιο κουράκι και να έχουν την ίδια δέσμευση με ε, την Φιλανδική Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τέλπο Κορφίλτα. Θα πρότεινα τώρα 1,5 λεπτά για τους σκιώδεις. Και επειδή Θέλουν και συντονιστέ συντονιστές και σκιώδει να τοποθετηθούν. Ε, παρακαλώ να τηρηθεί αυτό ο χρόνο. Ένα λεπτό, κύριε Μετσόλα. Ευχαριστώ, κύριε Τουκουράν. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που σα συναντάμε. Σα ευχαριστούμε πολύ για την ε, επαγγελματική και αποτελεσματική Προεδρία. Για το θέμα αυτό μπορώ να σα πω ότι το ΕΛΚ συμφωνεί με τι άλλε πολιτικέ ομάδε όσον αφορά τη συμμετοχή, την πλήρη συμμετοχή του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε και οι σκιώδεις εισηγητέ να ήταν ε, παρόντες σε αυτήν την άτυπη συνάντηση του προγεύματος, γιατί θα ήταν μια ευκαιρία να εκπροσωπηθούν όλες οι πολιτικές ομάδες και όλες οι πολιτικές απόψεις. Ως πολιτική ομάδα θεωρούμε πάντοτε ότι το κράτος δικαίου πρέπει να ε, εφαρμόζεται παντού και ότι οι αρχέ που κατοχυρώνονται στη συνθήκη θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστέ. Όμω βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν ε, μηχανισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίοι δεν είναι όσο αποτελεσματικοί θέλαμε ή ε, ανεπαρκείς ως προς την επίτευξη των στόχων για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να προβούμε σε, στη λήψη τιμωρητικών μέσων ποινών. Θέλουμε απλώς να ανταποκριθούμε σε αυτά που ε, περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ολοκληρωμένο και ανεξάρτητο μηχανισμό κράτους δικαίου που θα, που θα προσεγγίζει όλα τα κράτη-μέλη με αμεροληψία και ανεξαρτησία. Μόνο έτσι μπορούμε να ε, αποφύγουμε κατηγορίες ότι είμαστε ε, μεροληπτικοί εναντίον συγκεκριμένων χωρών. Χρειάζεται λοιπόν ίδιοι, ίσοι κανόνες. Ε, και βλέπω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να αλλάζει άποψη ανάλογα με το ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Αυτό το είδαμε τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα έντονα εδώ στο Κοινοβούλιο. Η κυρία Τκρούντεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ. Περάσαν τα χρόνια και ξεκίνησε μια νέα θητεία για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ενώ διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, ξεπερνάνε το ένα όριο μετά το άλλο. Ε, παραβιάζοντας το κράτος δικαίου, παραβιάζοντας ε, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, ε, προσπαθώντας να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον τύπο. Κάποιες φορές μάλιστα κανείς σχηματίζει την εικόνα ότι το κάνουν αυτό και απολαμβάνοντας πλήρη ασυλία. Πρόσφατα υπήρξαν επιθέσεις από την κυβέρνηση Ορμπάν εναντίον δικαστών, μέσων ενημέρωσης και τώρα πια και μέσω ε, εναντίον ε, θεσμών του πολιτισμού. Νομίζω ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να φιλοδοξεί μιλώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον νέο πρόεδρο του Συμβουλίου, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να φιλοδοξούν, να ε, επιμένουν ε, στο να λογοδοτούν όλοι εκείνοι που παραβιάζουν το κράτος δικαίου, να ενεργοποιούν το άρθρο 7 και να εφαρμόζουν μηχανισμούς για την αποτροπή πιθανών μελλοντικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είναι ε, τα πολιτικά κόμματα που κατέχουν ε, τις ε, κυβερνήσεις που πρέπει να επομίζονται και όχι οι λαοί που πρέπει να επομίζονται τις ε, επιπτώσεις για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Renew η κυρία Στρουγκάρου. Κάποιες σκέψεις για τα όσα συμβαίνουν ε, στην Ουγγαρία και με την Ουγγαρία. Όμως προτού σας παρουσιάσω αυτές τις σκέψεις μου θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση που νομίζω ότι είναι σημαντική. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε όλοι σε μια αμοιβαία συμφωνία, μια κοινή συμφωνία ότι υπό τον παρόντα, ισχύοντα κανόνα της ομοφωνίας του άρθρου 7 δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αγγίξουμε τον ε, Όρμπαν. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν μηχανισμό κράτους, του κράτους δικαίου που θα βάζει τέρμα σε τέτοιου είδους ιστορίες. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό για το κράτος δικαίου που θα είναι πολύ ισχυρό, με πολύ σαφείς και συγκεκριμένους κανόνες και δεν είμαι καν σίγουρη ότι και με έναν τέτοιο μηχανισμό όσο θα υπάρχει ο κανόνας για την ομοφωνία ότι θα, είναι, θα έχει κάποια αποτελεσματικότητα αυτός ο μηχανισμός. Δεύτερον, μόλις ε, γύρισα από μια διάσκεψη στη Βουδαπέστη για την ελευθερία του τύπου, η οποία πεθαίνει έναν αργό θάνατο στην Ουγγαρία. Και αυτό που ε, ένιωσα ε, στην αίθουσα που διεξαγόταν αυτή η διάσκεψη ήταν να ανατριχιάζει ο κόσμος όταν αναφερόταν το όνομα του Όρμπαν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια χώρα στην οποία ελέγχεται πλήρως ο τύπος. Και ξέρετε, ακούγονται ειδήσει ότι δεν υπάρχει ρωσική προπαγάνδα στην Ουγγαρία. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η προπαγάνδα του Όρμπαν είναι τόσο πανταχουπαρούσα και τόσο ισχυρή που δεν χρειάζεται τον Πούτιν. Πρόκειται για έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω, για το ποιος ε, κάνει καλύτερη προπαγάνδα. Επίσης, πρέπει επιτέλους να ενισχυθεί η διαφάνεια στο Συμβούλιο για τις ακροάσεις που κάνει, για την ομοθεσία που θεσπίζει. Γιατί αν δεν γίνει αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε tweets και διάφορες άλλες διαρροές με αυτόν τον τροπιαστικό τρόπο που διέρευσαν πληροφορίε από αυτή τη ε, συνάντηση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ ο Νίκολας Μπέι εκ μέρους του ID. Όχι δεν είναι εδώ. Άμα δεν είναι εδώ και δεν θέλει κανείς άλλος να μιλήσει εκ μέρους της πολιτικής ομάδας ID. Θα περάσουμε στην πολιτική ομάδα ECR. Η κυρία Βινιέσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Το άρθρο 7 έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό όπλο, μια, ένα μαστίγιο που χρησιμοποιείται εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων. Κάποιοι από εσά ε, φαίνεται να πιστεύετε ότι κάποιες κυβερνήσεις ε, δεν είναι αξιόπιστε επειδή δεν ακολουθούν τη δική σα πολιτική γραμμή. Προηγούμενοι ομιλητέ αναφέρθηκαν στα fake news, τι ψευδεί ειδήσει και την παραπληροφόρηση. Να σα υπενθυμίσω ότι κι εσείς πολύ συχνά συμβάλλετε σε αυτή την παραπληροφόρηση διότι επαναλαμβάνετε ειδήσει οι οποίε δεν έχουν επαληθευτεί και που απέχουν πάρα πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι είναι συμμαχία ε, κυρίαρχων εθνικών κρατών. Τα κράτη-μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις δικές τους ε, δημοκρατικές πλειοψηφίες και να σχηματίζουν μόνα τους τις κυβερνήσεις τους. Στην Αντίθετα με όλα αυτά όμως, αυτό που εσείς προσπαθείτε να κάνετε είναι να προσπαθείτε να ε, αναγκάζεται τα κράτη-μέλη να παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου. συνεχίζεται να δαιμονοποιείτε τον κύριο Όρμπαν και προσπαθώντας να μας πείσετε ότι οι Ούγγροι φοβούνται τον ε, πρωθυπουργό τους, τον Όρμπαν. Ε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να επαναλάβω ότι έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στην Ουγγαρία, η οποία θέλει να ε, λάβει υπόψη της κατά κύριο λόγο τις ανάγκες του λαού της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν είναι υπερκράτος, είναι μια συμμαχία εθνικών κρατών. Κυρία Μπιόρκ, είναι κάπου αλλού, δεν είναι εδώ. Η Κορνίλια Έρνστ εκ μέρους της Γκουε θα την αντικαταστήσει. Äh, Ακριβώς. Η Μάλιν Μπιόρκ είναι στην ε, Γενέβη για την συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία συμμετέχει να μην ξεχνάμε ποιο είναι το θέμα το οποίο συζητάμε. Αυτό που συζητάμε δεν είναι η αυτοδιάθεση κάποιου λαού ή κάποια πληθυσμιακή ομάδα, ούτε θέλουμε να καταστήλουμε τέτοια δικαιώματα, ούτε, για την, ούτε καν για την ανέρεση κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όχι, αυτό, που μιλάμε είναι, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι η βάση της δημοκρατίας. Γι' αυτόν τον σκοπό, γι' αυτόν τον λόγο πήγαν, βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους και στη χώρα τη δική μου το 89. Θέλαμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές για να υπάρξουν αυτές οι ελευθερίες για όλους. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μηχανισμό για το κράτος δικαίου, το είπε και συνάδελφος ο οποίος θα υπερβαίνει την ε, διαδικασία, την ε, διαδικασία ενεργοποίησης των διαδικασιών επί παραβάση και όλο αυτό το τσίρκο που μετά ακολουθεί. Συγγνώμη. Χρειαζόμαστε κάτι που θα υπερβαίνει όλα αυτά. Κάτι που θα ξεπερνάει την ε, αυταπάτη ότι μπαίνοντα κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελειώνουν τα, οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. State of play, λοιπόν. Ποια ήταν τα επιχειρήματα, τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη συνάντηση του Συμβουλίου, τι, τι ακριβώς καταφέρατε και τι δεν καταφέρατε, τι, τι, τι, βήματα σχεδιάζετε να κάνετε στο μέλλον. Γι' αυτά θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα. Όλοι οι συντονιστές πήραν το λόγο. Ή μάλλον όλοι συζήτησαν, όσοι από τους συντονιστές ζήτησαν το λόγο, θα τον πάρουν. 1,5 ε, λεπτό. Ε, η κυρία Σίπελ. Η κυρία Μετσόλα ήταν ε, σκιώδης. Αναφέρατε το εργαλείο για το κράτο δικαίου και τα προληπτικά μέτρα. Είπατε ότι 26 κράτη-μέλη συμφώνησαν. Αυτή την ερώτηση προ την Προεδρία του Συμβουλίου. Με εκπλήσατε λιγάκι. Μπορείτε να αξιολογήσετε ποια είναι αυτά τα εργαλεία, με τι μοιάζουν, τι κάνετε με αυτά. Δεύτερο σημείο. Ένα από του συναδέλφου το ανέφερε. Το νέο νόμο, όπως ο Υπουργό Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να αποφασίσει για τους διευθυντές των τοπικών θεάτρων. Αυτό έγινε μετά τις τελευταίες εκλογές. Αυτό συζητήθηκε την περασμένη Τρίτη στις Βρυξέλλες. Τους ρωτήσατε τι ακριβώς έγινε. Μιλήσατε επίσης για το γεγονός ότι τώρα το δικαίωμα της αντιπολίτευσης ε, στο Κοινοβούλιο δεν κατοχυρώνεται γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν πραγματική ομάδα. Ε, επίσης, δεν ήθελα να μπω στο ιστορικό των συζητήσεων για συστημική παραβίαση του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία στην Ουγγαρία, αλλά μου φαίνεται αστείο που ένας συνάδελφος λέει εδώ ότι πάντα ήταν ε, υπέρ του κράτους δικαίου και τώρα ε, εντυπωσιάζεται που κάποια κράτη-μέλη ε, αλλάζει άποψη επειδή αφορά την κυβέρνησή του. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την Ουγγαρία το 2009, πρέπει να σα υπενθυμίσω. Ήμουνα νέο μέλος, νέο, νέα βουλευτή και μας χρειάστηκε να ξοδέψουμε μια ολόκληρη κοινοβουλευτική θητεία. Την, πήραμε την απόφαση μόνη στην περασμένη κοινοβουλευτική θητεία για να βρούμε τελικά την απαραίτητη πλειοψηφία για να ομολογήσουμε ότι υπάρχει παραβίαση του κράτου δικαίου. Και αυτό γιατί εξαιτία μια ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο, μια πολιτική ομάδα. Και τώρα από το Ρηνιού η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα τη Φιλανδική Προεδρία, την κυρία Τουπουράινεν κυρίω. Ξέρω ότι σα απασχολεί πολύ αυτό το θέμα, έχετε δουλέψει πάρα πολύ από αυτού. Όμω πρέπει να καταλήξω συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα παρά τι προσπάθειε σα. Μπλα μπλα, αλλά δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Στο μεταξύ, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα βιάζονται και σκοτώνονται. Και τα κράτη-μέλη δεν κουνάν το δαχτυλάκι τους, απλώς παρίστανται στο φαινόμενο του βιασμού. Χαιρετίζω τις καλές σας προσπάθειες, αλλά η δημοκρατία πεθαίνει στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Υπάρχει απίστευτο απίθανος αυταρχισμό αυταρχισμός και από πίσω κρύβεται απίστευτη διαφθορά των ηγετών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το Συμβούλιο τι κάνει? Τίποτα. Ζητάμε από το Συμβούλιο να συζητήσει την κατάσταση στη Μάλτα. Όταν συναντήθηκαν ε, στη Σύνοδο Κορυφή την περασμένη εβδομάδα, συζήτησαν τη Μάλτα. Τίποτα. Ούτε κουβέντα. Στο μεταξύ, η αρρώστια απλώνεται. Το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ε, διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί χωρίς δημοκρατία, χωρίς κράτος δικαίου, χωρίς θεμελιώδη δικαιώματα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Ελπίζω οι συνάδελφοί σας επίσης επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνε σου για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Γιατί όταν ακούω τον Ολλανδό Υπουργό που λέει «Ναι, αυτά που συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες ήταν ησυχητικά». Αλλά είναι, ξέρετε, εθνικό θέμα. Όχι, κυρίε και κύριοι, δεν είναι εθνικό θέμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωσή μα. Και είναι και η ώρα το Συμβούλιο να αναλάβει τι ευθύνε του για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Να σταματήσει το μπλα μπλα για τον εθνικισμό, εθνικισμό και την εθνική κυριαρχία. Τώρα είναι η ώρα το Συμβούλιο να κάνει κάτι. Τώρα, εδώ και τώρα. I know we are confusing. Um, and I'm, also very happy that... Χαίρομαι που ήρθε εδώ, ήρθατε εδώ, κυρία Υπουργέ. Θα διαφωνήσω με το εξή. Με το εξής. Εγώ δεν έχω τόση εμπιστοσύνη όσο εσείς. Έχω και περάσει χρόνος και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα οδηγό για το πώς ε, θα, τα αυταρχικά καθεστώτα θα βαφτίσουν το καθεστώς, ας πούμε, δημοκρατία. Ε, έχουν, ε, απειλούν ας πούμε τους διαφορετικούς μειονότητες, τις διαφορετικές μειονότητες, ε, επιτίθενται στην κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών λένε ότι τις, τους απειλούν αυτές οι οργανώσεις, αλλά στην πραγματικότητα αποσταθεροποιούν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Επιτίθενται και στον πολιτισμό, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα κτλ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονό ότι αυτό δεν γίνεται μόνο σε ένα κράτο μέλο πια. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνονται αρκετά. Σα καλώ, σα κάνω έκκληση να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που έχει το Συμβούλιο για να γίνει κάτι. Ένα που δεν αναφέρθηκε είναι η συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και την αιρεσιμότητα. Να πείτε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να δημιουργείτε αυτό το αυταρχικό σα ολοκληρωτικό καθεστώ και να το παγιοποιήσετε και να το εδραιώσετε και να το προχωρήσετε. Όχι. Το Συμβούλιο πρέπει να, είναι στο πλευρό, στο πλευρό μας σε αυτό το θέμα. Thank you for be Mr. Ο κύριος Γιάκη είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Είναι μια συζήτηση που τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστηκαν πολλές φωνές που λένε θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτή η παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Έγινε πολλής λόγος ε, για τις ε, τεχνικές συνεδριάσεις, για τη ε, σημασία της ελευθεροτυπίας του κράτους δικαίου. Συμφωνώ και εγώ για ελευθερία των πανεπιστημίων, συμφωνώ. Όμως, το ερώτημα είναι πού παραβιάζεται το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Δεν είπε κανείς κάτι για αυτό, για να δούμε κατά πόσο να ευσταθούν ή όχι τα επιχειρήματα. Η κατάσταση επιδεινώνεται, λέτε, και τιμωρείται, τιμωρείται, τιμωρείται τη χώρα. Όμως, σας ζητώ όταν εγκαλείτε με τόσο σοβαρές κατηγορίες να μπορείτε και να τις επαληθεύσετε. Το πιο ενδιαφέρον επιχείρημα ήταν μίας ε, βουλευτού που είπε ότι τρομοκρατούνταν ακούγοντας ε, το όνομα του Όρμπαν. Μα πώς τρομοκρατούνται οι Ούγγροι και τον εκλέγουν τέσσερις φορές με τέτοια τεράστια πλειοψηφία. Το δικό σας κόμμα αγαπητοί συνάδελφοι. Ούτε στον ύπνο του δεν θα δει τέτοια αποτελέσματα. Αν είναι έτσι τότε να τρομοκρατήσετε, να τρομοκρατείτε και εσείς τους ψηφοφόρους όταν μιλάμε για παραβίαση του κράτους δικαίου. Ποια είναι αυτή η παραβίαση. Πριν ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, να ολοκληρώσουμε με όσους αδέλφους για ένα λεπτό καθένας θέλουν να κάνουν σύντομες ερωτήσεις. Insert. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Υπουργό ε, συγγνώμη, του Πουράινεν. Και σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας ε, το τελευταίο εξάμεινο. Σε συνέχεια των ερωτήσεων των συναδέλφων. Τα ρωτήσω και εγώ, τι μελγενέστε. Υπάρχουν παραβιάσεις. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν να το παραδεχτούν. ότι υπάρχει πολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος ε, στην Πόλωνη κτλ. Ξέρουμε όμως ότι αυτά είναι πραγματικότητα και για την Πολωνία. Είναι και απόφαση ε, να υπάρξει πολιτικοποίηση με νόμο. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Τι μέλη Πρόοδος υπάρχει. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα. για το τι μπορεί να γίνει προληπτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούγοντας τις ε, παρεμβάσεις, έχω την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με αριστερούς ιεροξεταστές. Είναι αδιανόητα τα πράγματα που ακούγονται από ανθρώπους που ε, περνούνται και για σοβαροί. Στην, ε, στην Ουγγαρία, λοιπόν, ε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πολιτικής επίθεση και πρόκειται για ένα κυνήγι μαγισσών στην πραγματικότητα. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες που τη απευθύνονται και έχει πάντοτε δηλώσει ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο. Δεν πρόκειται για διαδικασία η οποία ε, βασίζεται σε νομικά εργαλεία. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση για να επικριθεί η Ουγγρική κυβέρνηση για τα, χριστιανικέ. χριστιανικές ε, συντηρητικές αξίες της και για την στάση της απέναντι στην ε, ε μετανάστευση. Το πραγματικό θέμα που θα πρέπει να συζητάμε θα, ε, πρέπει να είναι η Μάλτα και η δολοφονία μιας δημοσιογράφου που μάλιστα θα συζητούνταν στην, στην Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα αλλά τελικά δεν θα συζητηθεί. Ναι, συζητάμε την Ουγγαρία λέει ο Πρόεδρος, έχουμε όμως και ένα σημείο για την Πολωνία και ένα σημείο για την Μάλτα. Απλά περιμένετε και θα δείτε. Η κυρία Τόναθ. Ευχαριστώ. Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 7 ως έσχατο μέσο μιας μεγάλης λίστας μέτρων εναντίον της Ουγγρικής κυβέρνησης που παραβιάζει το κράτος δικαίου. Δυστυχώ όμως τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Όρμπαν τελικά μόνο τον ενθαρρύνουν και τον παροτρύνουν να συνεχίσει στην ίδια οδό. Όπως ακούσαμε τώρα για τον διορισμό των διευθυντών των θεάτρων ή και την επιβολή κυρώσεων ακόμη και εναντίον βουλευτών. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να αναλυθούν αφού διαπιστώνουμε πια ότι η συνεργασία αντί να βελτιώνει τα πράγματα τελικά ενθαρρύνει την Ουγγρική κυβέρνηση να συνεχίζει και να εμβαθύνει την, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια ε, πλειοψηφία ε, γύρω από την πρόταση να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη διαφάνεια. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα στο Συμβούλιο, προς το Συμβούλιο. Ε, το οποίο είχα απευθύνει και το Σεπτέμβριο σε ακρόαση, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η Ουγγρική κυβέρνηση ζήτησε να γίνει μια τέτοια ακρόαση δημόσια ή ήταν απλά ε, μια κίνηση δημοσίων σχέσεων της Ουγγρικής κυβέρνησης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολλοί θεώρησαν ότι η έναρξη αυτής της διαδικασίας του άρθρου 7 θα ε, έβαζε μυαλό στον ε, κύριο Όρμπαν. Το αντίθετο έχει συμβεί. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ε, τον τελευταίο χρόνο, ιδίω μετά τις τοπικές εκλογές, όπου και οι τρεις τοπικές περιφέρειες, βιβλιοπολία, ακόμη και θέατρα έχουν γίνει στόχοι της κυβέρνησης του Φιντές. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι οι χριστιανοδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ούγγροι, επιμένουν ε, διαρκώς ότι το κράτος δικαίου είναι μία από τις βασικότερες χριστιανικές αξίες. Ελπίζω τους επόμενους μήνες να, συστοιχήσουν, να αντιστοιχίσουν μάλλον τα λόγια τους με τις πράξεις τους. Ότι δεν είναι δυνατόν η χριστιανοδημοκρατία να ταυτίζεται με τις ενέργειες και τις ε, πράξεις της κυβέρνησης Όρμπαν. Θα μιλήσω σλοβακικά. Ευχαριστώ. Πριν από ακριβώ δύο μήνε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας για τις παρεμβάσεις στις εκλογές. Οποιοςδήποτε λοιπόν λέει το αντίθετο, κατηγορείται ως προπαγανδιστής. Όμως όταν κάποιος αναφέρει τον Σόρος, τότε αμέσως κατηγορείται ως κάποιος που διασπείρει συνωμοσίες. Τελικά διαπιστώσαμε ότι αυτή, αυτό το πανεπιστήμιο που πήγε, να, κλείσει, να ανοίξει ο Σόρος και να κλείσει ο Ορμπάν τελικά δεν ήταν και πολύ πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γερμανικά. Ετέθηκαν πάρα πολλά ουσιώδη και σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να ε, ε, διερευνήσουμε και που η απάντηση που θα δώσουμε σε αυτά τα ερωτήματα βεβαίως θα επηρεάσει ε, σε μεγάλο βαθμό και συστηματικά την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η συζήτηση αυτή είναι και πολιτική αλλά και τεχνική. Τι εννοώ με αυτό. Πώς μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες πόσο σημαντικές είναι οι αρχές του κράτους δικαίου για την υπεράσπιση και την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διότι πράγματι ούτε στην Πολωνία ούτε στην Ουγγαρία έφτασαν στην κυβέρνηση αυτά τα κόμματα με πραξικοπήματα. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτούς τους αφηρημένους όρους του κράτους δικαίου να τους μετουσιώσουμε σε πραγματικά στοιχεία για τους πολίτες ώστε να μπορούν απτός να καταλάβουν τι εννοούμε. Υπάρχουν σκέψεις σχετικές στο Συμβούλιο. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά μέτρα για να, σπα... για να σταματήσουμε τη διάλυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η προστασία της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου είναι ε, τόσο σημαντικά. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μόνο στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ό,τι οι αρμοδιότητες έχουν. Έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 259. Είναι σπάνια, σπάνια χρησιμοποιείται για θέματα κράτους δικαίου. Γιατί ε, είναι κρίμα πάντως να αφήσουμε το πράγμα έτσι χωρί να κάνουμε τίποτα. Αν υπάρχει ένα πραγματικό συνασπισμό, κάτι μπορεί να γίνει. Ποια είναι η θέση τη Φιλανδική προεδρία, Έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάμε για την Ουγγαρία βεβαίω. Το πρόβλημα είναι με την Ουγγαρία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εναντίον τη Πολωνία όμω. Διερωτώ με. Υπάρχει στην ατζέντα του Συμβουλίου και των κρατών μέλων να κάνουν κάτι τέτοιο δυνάμει του 259. Ευχαριστώ. Λέει ο κ. Λαγκοντίνσκι, τρία σημεία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της αυτοθυματοποίησης. Όλες αυτούς τους χειρισμούς που ακούμε, εσείς πώς τους αντιμετωπίσετε στη συζήτηση που κάνετε με τις κυβερνήσεις. Η αοριστία της έννοιας αυτής του κράτους δικαίου είναι κάτι που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα. Ε, υπάρχει έλλειψη... Ε, λένε οι επικριτέ του κράτου δικαίου ότι είναι κάτι πολύ αόριστο. Αλλά υπάρχει τώρα νομολογία. Δεν είναι τόσο αόριστο πια. Έπειτα, μάλλον είναι η τελευταία σα φορά εδώ. Τι συμβουλή θα μα δώσετε μετά από την ε, διαδικασία που χρησιμοποίησατε και την εμπειρία που έχετε αποκοπήσει, Πώ μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτό το μηχανισμό για το κράτο δικαίου, κατά την απόψή σα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν μίλησε. Κυρία Σμέκα, μέσα σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, ναι, βεβαίω. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας, ε, για τη δουλειά που κάνετε για το κράτος δικαίου τους τελευταίους έξι μήνες. Θέλω να διευκρινίσω το εξή. Γιατί είμαι και εισηγητή ε, του Κοινοβουλίου για αυτό το νέο μηχανισμό κράτου δικαίου, δημοκρατία και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και χαίρομαι που πολλοί συνάδελφοι είναι υπέρ αυτή τη ιδέα. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια αμερόληπτη αξιολόγηση με βάση ξεκάθαρα κριτήρια που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Θέλω να πω ότι αυτό όμω δεν είναι υποκατάστατο του, της διαδικασίας του άρθρου 7 που έχει ξεκινήσει εναντίον της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία. Και μία σύντομη ερώτηση προς την Υπουργό. Είναι πιθανό τώρα στο κλείσιμο της Προεδρίας ο επόμενος ετήσιος διάλογος για το κράτος ε, δικαίου στο Συμβούλιο να γίνεται με βάση την έκθεση της Κομισιόν. Είχε ξεκαθαριστεί αυτό, είναι δεδομένο. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρο, πρόεδρος, άνευ μικροφώνου. Λοιπόν, έχει μείνει λίγος χρόνος γιατί προβλεπόταν μέχρι τις 10 και μισή να συνεχιστεί η συζήτηση, άρα έχουμε χρόνο και μπορείτε να κάνετε εσείς κάποια σχόλια τώρα. Δεν θα είναι ικανοποιημένοι όλοι, γιατί θα σας δώσω πέντε λεπτά ότι θα μπορείτε να απαντήσετε σε όλους, αλλά ούτως ή άλλως δεν κλείνει εδώ το θέμα. Είναι πολύ βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΑ αυτά τα θέματα. Κάντε λοιπόν τις δικές σας δηλώσεις, 5-7 λεπτά μετά εσείς, ε, πρώτα έσως ο Επίτροπος ε, Ρεντέρς και μετά η κυρία του Πουράινεν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσήλωσή σας στο κράτος δικαίου, γιατί και από τις προηγούμενες συζητήσεις βλέπω ότι αυτή η όλη διαδικασία ξεκίνησε από το Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έχοντα ε, την καλή συμμετοχή και των θεσμικών οργάνων. Άρα, παρόντου και το Κοινοβούλιο, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα έχουν υποθεί. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μα πάνω στο άρθρο 7 και με την Κροατική Προεδρία. Ε, ξεκινήσαμε και με ε, τη Φιλανδική Προεδρία και θα συνεχίσουμε την Κροατική και έχουμε καλή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Υπάρχει αυτή η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος δικαστών. Υπάρχουν και άλλες ε, πρόσφατες εξελίξεις με νέα νομοθεσία που είχε να κάνει με την εξαρτησία των δικαστών στην Ουγγαρία. Άρα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, στην εργαλειοθήκη μας έχουμε και άλλα εργαλεία. Και επαναλαμβάνω ότι η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η θα συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάση όταν αυτό είναι αναγκαίο με την Ουγγαρία για το δεύτερο βάθμο εκπαίδευση. Περιμένουμε την απόφαση του καστηρίου. Το ίδιο με την Πολωνία. Και το τρίτο στοιχείο, φυσικά και θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλος. Θα είναι δική μου αρμοδιότητα στην Κομισιόν να οργανώσω τη, το νέο μηχανισμό με όλα τα κράτη-μέλη ακρίτως θα συζητήσουμε. Θα είναι ένας νέος μηχανισμός. Χωρίς όμως να εγκαταληφθεί η διαδικασία του άρθρου Έχουμε απλά ένα νέο εργαλείο που προστίθεται στη φαρέτρα μας. Και τέλος, η, η χρηματοδότηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και η αιρεσιμότητα στο πιδελταπή είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες συνέπειες τέτοιων παραβιάσεων, γιατί σαν είναι συστηματικές αυτές παραβιάσεις του κράτου δικαίου. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, γιατί θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, συνεχίζει η διαδικασία των τρεπτά, αλλά θα συνεχίσουμε και με άλλα εργαλεία τα οποία θα προσθέσουμε στην εργαλειοθήκη. μα. ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ γιατί ήσασταν ε, σύντομος και σαφής. Ε, κυρία Τουπουράινεν, εσείς το έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ για τι ε, πολύ σημαντικέ ουσιώδει παρεμβάσει σα. Δυστυχώ δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν, γιατί ήταν πολλέ οι παρεμβάσει. Όμω σα διαβεβαιώ ότι σημείωσα όλα αυτά που είπατε, όλε τι παρατηρήσει σα και βεβαίω δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Να ξεκινήσω με την παρά Τήρηση της κυρίας Δελβός για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ακροάσεις του άρθρου 7 στο Συμβούλιο. Ναι, πράγματι συζητήθηκε δεόντως αυτό στην προετοιμασία των τυπικών διαδικασιών που προηγήθηκαν των ακρεώσεων. Αυτές οι τυπικές διαδικασίες ε, διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τη νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου. Και το άρθρο 7 ε, προβλέπει το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί και δίνει τη συγκατάθεσή του. Δεν προβλέπει κάποια μεγαλύτερη, κάποιο μεγαλύτερο ρόλο του άρθρου 7 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενημερώνεται το Συμβούλιο για τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα πρέπει να ενισχύεται η συμμετοχή του, όπως ήταν και η δική σας πρωτοβουλία. Γι' αυτό και στη διάρκεια της Προεδρίας μου μας ε, έκανα ό,τι περνούσε από τα χέρια μου σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς πράγματι ε, υπήρξε αυτό το ατυχές γεγονός με το Twitter στην ε, διάρκεια της τελευταίας ε, ακρόασης του άρθρου 7 στο Συμβούλιο. Ήταν πραγματικά κάτι αξιολύπητο και ζήτησα Μέσω εξήγηση από την Ουγγρική Αντιπροσωπεία για τη συμπεριφορά του και μάλιστα έλαβα τάχιστα και μια απάντηση από την Ουγγρική Κυβέρνηση ε, ε, η οποία ήταν όμω και ανεπαρκής, ε, πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, περιλάμβανε αμφιλεγόμενες υπόνοιες εναντίον του Συμβουλίου και γι' αυτό και ζήτησα από το ΚΟΡΕΠΕΡ, το Σώμα των Μονίμων Αντιπροσωπιών, να συζητήσει το θέμα αυτό. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί και νομίζω ότι σήμερα πια ε, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι έχουν συζητήσει πλέον το θέμα και θα το διευθετήσουν με οριστικό τρόπο ε, και βεβαίως θα απαντήσουμε και στις κατηγορίες που απίφθινε η Ουγγρική κυβέρνηση στην Προεδρία του Συμβουλίου με τον ε, δέοντα τρόπο. Βεβαίω, το να στέλνει κανεί tweets σε διάρκεια μια τέτοια ακροαση δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν μα. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στα εργαλεία και στου μηχανισμού που έχουμε στην διάθεσή μα στον τομέα του κράτου δικαίου. Εμεί ω Προεδρία κάναμε ό,τι μπορούσαμε και σημειώσαμε πρόοδο σε τρει άξονε. Πρώτον, ξεκινήσαμε τι ακροασει του άρθρου 7 με την Ουγγαρία. Νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μα να το κάνουμε αυτό. Κάναμε αυτό ακριβώ που περιμένατε από εμά και δεν ήταν καθόλου εύκολο πρέπει να σα πω. Υπήρχαν και κάποια σχόλια ότι δεν ήταν και καθόλου ευχάριστη όλη η εμπειρία. Όμως με την δική σας πρωτοβουλία και πρόταση θεωρήσαμε ότι ήταν πλέον καιρός να ξεκινήσουμε. Επίση, συνεχίσαμε τις διαδικασίε εναντίον της Πολωνίας. Είχαμε κάποιου απολογισμού και κάποιε ενημερώσεις και θα, συνεχίσουμε, θα συνεχίσετε βεβαίω με αυτό το θέμα στη συνέχεια. Και διάλογος για το κράτος δικαίου. Υποβάλαμε συμπεράσματα ε, της Προεδρίας για τον απολογισμό και την αξιολόγηση του διαλόγου για το, το, για το κράτος δικαίου και χαίρομαι πάρα πολύ που από εδώ και πέρα στο μέλλον θα υπάρχει peer review, ε, εξέταση ομοτήμων, ε, αξιολόγηση ομοτήμων που θα βασίζεται πλέον σε αυτή τη μελέτη και ελπίζω ότι και στο μέλλον αυτή η διαδικασία θα ακολουθεί και από την Κροατική και από την Γερμανική Προεδρία. Και τέλος, υπάρχει η αιρεσιμότητα του ΠΔΠ. Για μας ως Προεδρία, όταν εκδώσαμε τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές μας για τη διαπραγμάτευση εν ώψη του ΠΔΠ, είχαμε πει ναι για αιρεσιμότητα και για κράτος δικαίου. Όταν κάποιος λοιπόν ε, θα διαπιστώνεται ότι κάποια κυβέρνηση παραβιάζει αρχές του κράτους δικαίου μπορούν να παγώνουν τα κονδύλια που κατευθύνονται προς αυτήν. Θα πει κάποιος ότι θα πρέπει να έχουμε αποτρεπτικά εργαλεία. Ε, η αιρεσιμότητα είναι ακριβώς αυτό το εργαλείο που χρειαζόμαστε και που θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Κυρία Βυσνιέσκα. Ναι, η Ουγγρική κυβέρνηση και η Πολωνική κυβέρνηση προφανώ και έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Δεν μπορεί κανεί να πει ότι δεν είναι δημοκρατικέ κυβερνήσει. Όμω, όταν υπάρχει κράτο μέλο με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, όλοι δεσμεύονται από του ίδιου κανόνε. Και σε αυτό επιμένουμε εμεί. Όταν μιλάμε για το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε για τη συμπεριφορά μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, ούτε για τις πολιτικές απόψεις ή τις ηθικές απόψεις που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση. Μιλάμε για την τήρηση των νομικών κανόνων που κατοχυρώνονται στη συνθήκη. Το άρθρο 2 λέει, αναφέρει ότι το κράτος δικαίου είναι θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είμαστε τόσο αμήλικτοι με αυτό το θέμα και άτεγκτοι. Και τέλος, με ρωτήσατε τι συμβουλές έχω. Υπάρχει μια φιλανδική λέξη «σίσου» που σημαίνει ανθεκτικότητα, αντοχή. Οπότε δεν παραδεινόμαστε, συνεχίζουμε και το ίδιο καλούμε να κάνουν και η Κροατική Προεδρία και όλες οι επόμενες προεδρίες που επίκυνται. Αυτή είναι η κληρονομιά μας, η παρακαταθήκη μας. So good to see you with so much Χαιρόμαστε που έχετε τόσο πολύ σίσου και τόσο πολύ ενέργεια. Συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα. Και εμείς συνεχίζουμε, χωρίς ανάπαυλα, για τη διαδικασία του άρθρου 7.1 σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει στην Πολωνία για το κράτο δικαίου. Το Κοινοβούλιο υιοθώθησε διάφορα ψηφίσματα, κυρίω εκείνο που υιοθετήσαμε το Μάρτιο του 2018, που ήταν υπέρ τη ενεργοποίηση του άρθρου 7.1 τη διαδικασία αυτή εναντίον τη Πολωνία ξεκίνησε από την Κομισιόν με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα πήρατε και το προβάδισμα ε, με την ε, Ουγγαρία και με την Πολωνία. Ο προκάτοχός μου, ο Κλοντ Μωράες, ε, πήγε στην Βαρσοβία σε μια αποστολή της Λίμπε, μίλησε σε προσώπους κυβέρνησης, ε, στην, ε, με προσώπους του Πολωνικού Κοινοβουλίου, δικαστές, ε, δημοσιογράφους. Η αποστολή αυτή οργανώθηκε καθώς και μία ακρόαση από τη Λίμπε τον Νοέμβριο πέρυσι και βλέπουμε τι γίνεται ε, απειλές εναντίον των δικαστών, απειλές εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ Ανισχούμε πάρα πολύ για τις πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των δικαστών που επικρίνουν τις μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης. Περιμένουμε να ακούσουμε συγκεκριμένα στοιχεία από τους δύο μιλητές μας, από την ε, Υπουργό και τον Επίτροπο, για τα θέματα αυτά. Εγώ ήμουν εισηγητής για αυτό το θέμα. Σας καλώ όλους να κάνετε ό,τι μπορείτε για να συζητήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το σημείο τέτοια ώρα, τόσο αργά. Ας χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο το χρόνο. Σας δίνω το λόγο για 5 με 7 λεπτά για να παρουσιάσετε το πλαίσιο. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω το πώς έχει κατάσταση σε σχέση με την κατάσταση του στην Πολωνία στο πλαίσιο του 7 παράγραφος 1 και τη σχετική διαδικασία. Καταρχά, να σα υπενθυμίσω πω ε, είναι διαφορετική αυτή η διαδικασία σε σχέση με την Ουγγαρία σε δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το ξεκίνησε αυτή τη φορά η Κομισιόν. Και πριν ξεκινήσει επίσημα τη διαδικασία του άρθρου 7, Ευχαριστούμε για πρώτη φορά για την Πολωνία αυτό το πλαίσιο για το κράτος δικαίου. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πεδίο, το εύρος, είναι ε, λίγο πιο στενό, ε, ενώ για την Ουγγαρία 12 διαφορετικά θέματα καλύπτονται. Για την Πολωνία η κατάσταση μόνο ε, αφορά το δικαστικό σώμα. Όταν ξεκίνησε ε, στις αρχές Ιουλίου ε, η Προεδρία Ήδη ήταν σε πλήρη εξέλιξη δικασία για την Πολωνία. Τρει ακροάσει είχαν γίνει επί Αυστριακή Προεδρία. Και στη διάρκεια τη Φιλανδική Προεδρία, η δικασία για την Πολωνία ήταν στην ημερήσια διάταξη του Σύμφωνου Γενικών τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο και τι τρει φορέ ω state of play. Οι συζητήσεις αφορούσαν ε, τις αποφάσεις της πρόσφατες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ζητήματα τα οποία καρπτονται από τη διαδικασία του άρθρου 7. Αποφάσεις που έδωσαν ε, σαφήνεια ε, και επέλυσαν κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα. Στη συνεδριά του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ημερώθηκε το Συμβούλιο για τις αποφάσεις, τι επιπτώσεις έχουν και ενημέρωση και για άλλες εξελίξεις σχέση με το δικαστικό σώμα στην Πολωνία. Η πολωνική κυβέρνηση φυσικά έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει και να δώσει πληροφορίες. Κατά την άποψή μου, επρόκειτο για χρήσιμες ανταλλαγές, μας επέτρεψαν να δούμε πιο καλά την εικόνα της κατάστασης στην Πολωνία. Αυτά αγαπητοί φίλοι και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ρέντρες για να σας πει περισσότερα για την ουσία. Ευχαριστώ και βέβαια παραμένω στη διάθεσή σας. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να σας εκφράσουμε την δική μας άποψη της Κομισιόν. Είχαμε την ευκαιρία με την κυρία Γιούροβα να ενημερώσω το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 10 Δεκεμβρίου για την κατάσταση στην Πολωνία. Να ξεκινήσουμε με τις ε, εξελίξεις ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 5 Νοεμβρίου το δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση σε μία από τις ε, περιπτώσεις παραβάση εναντίον της Πολωνίας σε ό,τι αφορά ε, τις αλλαγές που γίνονται στα τακτικά δικαστήρια. Οι δικαστές στηρίζουν την άποψη της Κομισιόν και αποφάσισαν ότι χαμηλώνοντας το σταξιωτικό όριο για τακτικά δικαστήρια και δίνοντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να παρατείνει την, την υπηρεσία τους, αφού φτάσουν στο συνταξιδοτικό όριο, παραβιάζεται η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ε, και το άρθρο 91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σημαντική απόφαση που δίνει και την νομική βάση για τους δικαστές που επηρεάζονται από το ε, εν λόγω νομοθέτημα να ζητήσουν ε, διόρθωση. Στις 19 Νοεμβρίου το δικαστήριο εξέδωσε μια νέα απόφαση, μια προδικαστική απόφαση σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του, της νέας ε, πειθαρχικής, ε, του νέου πειθαρχικού σώματος που πρόσφατα δημιουργήθηκε. Το δικαστήριο ζήτησε ότι το, είπε ότι το ανώτατο δικαστήριο της Πολωνίας πρέπει να αποφασίσει αν το νέο αυτό ε, πειθαρχικό σώμα είναι ανεξάρτητο και να δώσει διάφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση αυτή. Κυρίως το ανώτατο δικαστήριο έπρεπε να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του πειθαρχικού σώματος διορίζονται, ιδίως η επιλογή τους από το νέο Συμβούλιο Δικαιοσύνης που πρόσφατα δημιουργήθηκε. Το Ανώτατο Δικαστήριο έπρεπε να λάβει υπόψη ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου δικαστές εκλέγονται από το Κοινοβούλιο και όχι πια από τους ομοτήμους τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το Εθνικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντά του. Το Ανώτατο Δικαστήριο επίσης έπρεπε να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το πειθαρχικό σώμα αποτελείται μόνο από νεοδιοριστέντες δικαστές και ο... έχει μεγάλο βαθμό εξαρτησίας ε, από το ανώτατο δικαστήριο. Με την προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το ανώτατο δικαστήριο της Πολωνίας υιοθέτησε την απόφασή του στις 5 Δεκεμβρίου και αποφάσισε ότι το πειθαρχικό σώμα αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ε, του ευρωπαϊκού δικαίου για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και επομένως δεν ε, την, δεν σέβεται το ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο. Το ανώτατο δικαστήριο είπε ότι το εθνικό δικαστήριο Εθνικό Συμβούλιο μάλλον Δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητο από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Ένα μήνυμα από τους διερμηνείς ότι πρέπει να διαβάσετε λιγάκι πιο αργά. Και επομένως το ανώτατο δικαστήριο με την απόφασή του τονίζει ότι η ερμηνεία του Ενωσιακού Δικαστηρίου στις 19, 19 Νοεμβρίου με την απόφαση είναι δεσμευτική για κάθε δημόσιο φορέα και δημόσια αρχή στην ε, Πολωνία. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις από τις πολωνικές κρατικές αρχές που επικρίνουν το, την απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου της Πολωνίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου σημαίνει ότι όλες οι κρατικές αρχές έχουν την ε, υποχρέωση να σέβονται τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ισχύει ακόμα και όταν αυτές οι αποφάσεις ε, ε εκδίδονται εφαρμόζοντας σε μια προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπως είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στην ομολογία του, η αρχή της πρωτοκαθεδρίας του ενωσιακού δικαίου ερμηνεύεται ως ε, νόμος που υπερισχύει σε σχέση με το εθνικό δίκαιο. Επομένως, ήγηκε η ώρα για τις πολιτικές αρχές να δείξουν τη δέσμευσή τους απέναντι στο κράτος δικαίου. Ε, υπήρχαν και άλλες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την απόφαση ε, του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 19 Νοεμβρίου. Ένα κατώτατο δικαστήριο προσπάθησε να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υπέστη πειθαρχικές διώξεις από ε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο εν λόγω δικαστής αυτού του δικαστηρίου απομακρύνθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχε ε, αποσπαστεί σε εκείνο το δικαστήριο ε, και απομακρύνθηκε από τη θέση του. Ο, πρόεδρος, ο δικαστής αυτής είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Κάτι που συνδέεται άμεσα. Στις 3 ε, Δεκεμβρίου ε, δημοσιεύθηκε μία δήλωση που επικρίνονται αυτές οι δικαστές που αμφισβήτησαν το καθεστώς άλλων δικαστών. Στην ίδια δήλωση η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης. Επίσης μαθαίνουμε ότι στις 4 Δεκεμβρίου το, το πειθαρχικό αυτό σώμα ξεκίνησε διαδικασίες εναντίον του Προέδρου της μεγαλύτερης οργάνωσης ε, δικαστών στην Πολωνία, τη Ζουστίσια. Ε, γιατί αμφισβήτησαν την απόφαση του Πειθαρχικού Σώματος και του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτές οι αντιδράσεις είναι κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ε, δημιουργήθηκε μια τέτοια κατάσταση στο, μεταξύ των δικαστών και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για την κατάσταση του κράτους δικαίου. Ε, επιπλέον, στις 12 ε, Δεκεμβρίου η πολωνική κυβέρνηση υπέβαλε ένα νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για νέα δικήματα που αφορούν το πειθαρχικό καθεστώς των δικαστών καθώς και τη διαδικασία για το διορισμό του νέου πρώτου Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η Κομισιόν αναλύει αυτή τη στιγμή το σχέδιο νόμου, το το νομοσχέδιο αυτό με βάση τι προποθέσει του ενωσιακού δικαίου σε ό,τι αφορά την εξαρτησία τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να σε ενημερώσω επίση για τη χρήση τη πειθαρχική διαδικασία εναντίον των δικαστών. Η Κομισιόν αποφάσισε στις 10 Οκτωβρίου του 2019 να παραπέμψει την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε διαδικασία παραβάση σε ό,τι αφορά το νέο πειθαρχικό καθεστώ. Σε ό,τι αφορά, η, μάλιστα η Κομισιόν θεωρεί ότι το νέο καθεστώς αυτό το πειθαρχικό δεν δίνει τις απαραίτητες εγγυήσει για την προστασία των, δικαστών από τον πολιτικό έλεγχο ε, με την επιφύλαξη αυτή, οι νέες πειθαρχικές διαδικασίες ξεκινούν εναντίον δικαστών. Σύντομα, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά άλλους ισχυρισμούς ότι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αλλάζει τη σύνθεση των ε, ομιλητών των ακροάσει με βάση πολιτικά κριτήρια. Στις 4 Δεκεμβρίου, δύο δικαστέ του δικαστηρίου δήλωσαν δημόσια ότι στην τρέχουσα κατάσταση το συνταγματικό δικαστήριο δεν μπορεί σε θέση να διασφαλίσει αποτελεσματικά το κράτο δικαίου στην Πολωνία. Επίση, η Κομισιό γνωρίζει ότι ο Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρος τη δικαιοσύνη σε διάφορε φάσει ε, είπαν ότι θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις της ε, δικαιοσύνης. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στον τομέα αυτό. Κλείνοντα, Πρόεδρε, λυπάμαι που οι εξελίξει του τελευταίου μήνα δείχνουν ότι η κατάσταση στην Πολωνία επιδεινώνεται έτσι περαιτέρω. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση και είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει με τις πολωνικές αρχές τα θέματα αυτά. Βεβαίως, είμαι στη διάθεσή σας να, κρατώ, να σας τηρώ ενήμερους και σας και το Κοινοβούλιο. Χρειάστηκε να μακρηγορήσω γιατί έπρεπε να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα θέματα ε, που έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν. Thank you so much for Ευχαριστώ για τις ε, σαφείς και τολμηρές θα έλεγα, δηλώσει σα. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ω εξή. Πρώτα, θα γίνει ένας ε, γύρος ε, τοποθετήσεων από τους συζητητέ, που τυχαίνει να είμαι εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και συνέχεια θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Αλλά υπάρχει και ένας κατάλογος ομιλητών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συντονίσω ε, τον ε, χρόνο ε, φαίνεται ότι μάλλον τελικά θα υπερβούμε λίγο το χρόνο της συνεδρίασής μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να επιτεχύνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται. Πρώτα απ' όλα, προφανώς σεβόμαστε πλήρως την Πολωνία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα μεγαλύτερα σε πληθυσμό. Οπότε με ανησυχία και προβληματισμό κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία δηλαδή τις πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πολιτικό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2015 ήδη, η τεχνητή μείωση, κάτι που δεν το λέει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η Επιτροπή της Βενετίας και άλλοι διεθνείς ε, οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τολμαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τεχνητή μείωση λοιπόν του ορίου συνταξιοδότησης των ε, ε, δικαστών κάτι που σταμάτησε μόνο μετά από παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να μπορούν να επιλέγονται δικαστές που θα είναι αφοσιωμένοι στην κυβέρνηση. Ο εναγκαλισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης με τον ε, Γενικό Εισαγγελέα και τις εισαγγελικές αρχές και το ζήτημα που σχετίζεται με το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικαστών, στο οποίο επίσης διορίζονται, τα, το, του τα μέλη επίσης διορίζονται από την κυβέρνηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη προδικαστικά για το Πειθαρχικό αυτό Συμβούλιο και τη συμπεριφορά του Συμβουλίου αυτού και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρήχε στο Πολυνικό Συνταγματικό Δικαστήριο ένα αναλυτικό πλαίσιο για να ελέγξει αν εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμυροληψία των δικαστικών αρχών όπως αυτή κατοχυρώνεται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι το Εθνικό Δικαστήριο δεν είναι επαρκώ ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Και το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στα όσα ορίζει το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Απευθύνα λοιπόν τρία ερωτήματα στην Κομισιόν, στα οποία νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε ο Επίτροπος τι θα κάνει η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει τις ανησυχητικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον πρωταρχικό ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνικού, που είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το ε, ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δεύτερον, ενημερωθήκαμε ότι μια ομάδα Πολωνών και διεθνών ακαδημαϊκών πανεπιστημιακών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνυπέγραψαν επιστολή αυτή την εβδομάδα που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητείται η Κομισιόν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ε, έκδοση ασφαλιστικών μέτρων προτού ε, ε μπορέσει η πολιτική κυβέρνηση να λάβει παθαρχικά μέτρα εναντίον δικαστών προτού βγει το, η οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα θέλαμε την άποψη της Κομισιόν από αυτού. Και τέλος, θέλουμε να μας πείτε ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί το επόμενο διάστημα όσον αφορά τα προβλήματα κράτου δικαίου στην Πολωνία. Και ιδίω όσον αφορά την ενεργοποίηση τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφο 1. Ο λόγο του σκιώδη των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος στους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. 1,5 λεπτό στους Σκιώδης και 1 λεπτό τον πολύ σε κάθε μέλος της Επιτροπής. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε ότι καταφέρθηκε ακόμα ένα πλήγμα με το νέο πειθαρχικό καθεστώς κατά του κράτους και στην Πολωνία και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχούμε εδώ και καιρό με τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις ε, που εφαρμόζονται και που τελικά εδραιώνουν τον κρατικό έλεγχο, αποδυναμώνουν τους θεσμούς ε, που στόχο ήταν να ε, αποτελούν ένα θεσμικό αντίβαρο. Είδαμε να μην υπάρχει προθυμία από την πολιτική κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο να λάβει υπόψη τη συστάση επιτροπή, το πειθαρχικό πλαίσιο ουσιαστικά δεν είναι τα χέρια των δικαστών και τιμωρεί όσους έχουν ασκήσει κριτική ε, στην επιρροή που ασκεί η κυβέρνηση στα δικαστήρια. Υπάρχουν πειθαρχικές έρευνες, επιβολή κυρώσεων με βάση αποφάσεις των δικαστών ακόμη και όταν ασκούν το δικαίωμα προδικαστικού ερωτήματος που καταβάλλεται στην, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ένωσης. Άρα δεν υπάρχουν τα πάντα αντίβαρα που να εξασφαλίζουν ότι αυτές οι πειθαρχικέ διαδικασίες θα είναι ε, δίκαιες και δεν θα υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Μιλήσατε και για το τελευταίο νομοσχέδιο τη προηγούμενη εβδομάδα ε, με στόχο ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δικαστών. Απαράδεκτο το θεωρούμε. Γι' αυτό χαιρόμαστε κύριε Ρέιντερς που είπατε ότι δεσμεύεστε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου να είναι σεβαστά. Το είπαμε και στην προηγούμενη ε, συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητή. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που μας ε, εξήγησε την περίπτωση της, Ουγγαρή, της Πολωνίας ε, που είναι ανησυχητική και καλά κάνει και ανησυχεί με τις εξέλιξεις του τελευταίου μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατάσταση κατάσταση μέρα με τη μέρα θα έλεγα εγώ επιδεινώνεται. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δικαστές και συγκελείς από την Πολωνία που μας είπαν απίστευτα πράγματα για τις διώξεις που υφίστανται αυτοί και οι οικογένειές τους. Τους παρενοχλούν ήδη οργανωμένες εκστρατείες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, εφαρμόζονται σε βάρος τους. Και υπάρχει και αυτός ο νέος νόμος, όλοι αναφερθήκατε σε αυτόν, που κυριολεκτικά επιτρέψει το κυβερνών κόμμα να απολύει, να καθαίρει δικασίε που θέλουν να εφαρμόσουν αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται κάτι εντελώ ε, ε, καινοφανές ε, που κάνει τα πράγματα πολύ σοβαρά. Και η ουσία του ερωτήματό μου, το κάνατε κι εσείς αυτό το ερώτημα, ποια είναι τα προσωρινά μέτρα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση για τη νέα πειθαρχική διαδικασία, το φορέα αυτό ε, στην Πολωνία. Μήπως θα έπρεπε να προτείνουμε προσωρινά μέτρα, ασφαλιστικά δηλαδή, μέτρα για να συγκρατηθεί η ζημία που θα δημιουργήσει η δημιουργία αυτού, που, η έναρξη ε, αυτού του νέου δικαστικού πειθαρχικού σώματος. Ευχαριστώ και από τους Πρασίνους για 1,5 λεπτό. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να βρούμε περισσότερο χρόνο για αυτή τη συζήτηση, ίσως να οργανώσουμε τον Επίτροπο και τη Νέα Προεδρία μια άλλη συζήτηση, για να μην τα συζητάμε 10.30 το βράδυ, αλλά με το φως της ημέρας, για να είναι και άλλοι παρόντες. Πολλά υπόθηκαν και εσείς πολύ εύκολα μας παρουσιάσετε την κατάσταση ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και τη διάκριση εξουσιών. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι διαφορετικό που είναι το παιδί εφαρμογή τη καθέση των τριφτά σε βάση Πολωνία. Γιατί πράγματι το θέμα είναι η δικαστική μεταρρύθμιση και η ανεξαρτησία των δικαστών. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε και πιο πέρα. Αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα ψήφισμα με το οποίο λέμε ότι και η κατάσταση των θεμελιδών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη προσοχή και έχετε ίσω ακούσει τι δηλώσει για λεγόμενες ε, ε, απαλλαγμένες από ΛΟΑΤΚΙ ζώνες. Και όλες αυτές οι εξελίξεις πραγματικά είναι λόγοι σοβαρής ανησυχίας. Ε, οι μειονότητες ε, διώκονται, ιδίω οι ΛΟΑΤΚΙ. Και εμείς στην Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο που θέλουμε να περιφρονήσουμε τα δικαιώματα των δικαιωμάτων θα πρέπει να το κάνουμε και στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αθροεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να σας ηρεμήσω και να σας καθησυχάσω, δεν θα σταματήσουμε εδώ να συζητάμε το κράτο δικαίου και την καταστασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουν και άλλε συζητήσεις αρχές του 2020. Απλώς αυτή είναι η τελευταία συζήτηση για το 19. Έτσι. Τώρα. Ο σκιώδη του ID δεν είναι εδώ. Ο κύριο Μπέι δεν είναι εδώ. Άρα πάμε στο σκιώδη του ECR. Ο κύριο Μπρουτζίνσκι. Είναι εδώ. Το αντικαθιστάτε εσεί βεβαίω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, Επίτροπε, δεν έχουμε χρόνο να διορθώσουμε όλες τις ανοησίες που ακούσαμε. Είπατε ότι το πειθαρχικό σώμα δεν διορίζεται από δικαστέ. Διορίζεται από το Κοινοβούλιο. Όχι. Όχι διορίζεται από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης που απαρτίζεται από δικαστές. Σε ό,τι αφορά το δικαστήριο τώρα. Να διορθώσουμε το εξής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάλεσε το Πολωνικό Δικαστήριο να εξετάσει τη διαδικασία διορισμού των δικαστών. Το άρθρο 135 δεν επιτρέπει στους μεμονωμένους δικαστές να αμφισβητούν το καθεστώς των άλλων δικαστών. Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δικαστήριο, κανένας δεν έχει διωχθεί. Απλώς η θητεία κάποιων δικαστών έληξε. Εσείς κάνετε σοβαρότερες κατηγορίες. Ασκείτε ε, ε, και εξαπολύτε διάφορες κατηγορίες δεξιά και αριστερά. Σας παρακαλώ, είστε επαγγελματικός, έτσι μεταρρυθμι... Ε, αξιολογείται τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην Πολωνία με βάση κάποια σλόγγαν. Ακούτε μόνο τη μία σκοπιά, τη μία πλευρά. Μόνο κάποια επιχειρήματα. Δίνετε την εντύπωση ότι γνωρίζετε περισσότερα από, την, ε, από τους πολίτες μας για την Πολωνία. Τι ξέρουν οι Πολωνοί πολίτες. Ξέρουν αυτά για να επανεκλέξουν την ίδια κυβέρνηση. Τώρα, αυτά ήθελα να πω για τη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης. Θα ήθελα όμως να συνεχίσω να μιλάω αργότερα και ω συντονιστή. Θέλετε να μιλήσετε ως κοιόδης τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Αν με ηρεμία κοιτάξει τη συνολική εικόνα κανείς, διαπιστώνει ότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία είναι τόσο βαθιές πλέον που βλάπτουν μακροπρόθεσμα τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας. Και είναι πραγματικά ευτυχέ το γεγονό ότι τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, βγαίνουν στον δρόμο και δείχνουν την αλληλεγγύη τους στου συμπολίτε τους. Και μου είναι δύσκολο να μιλάω για όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι γειτονική χώρα η Πολωνία. Λίγα χιλιόμετρα από τα γερμανοπολωνικά σύνορα ζω εγώ. Έχουμε πολλές επαφές και με ανθρώπους και με δημάρχους και με οργανώσεις και αντιλαμβάνομαι κι εγώ και ότι υπάρχουν πιέσεις που ασκούνται σε αυτή τη χώρα. Και το λέω με πόνο ψυχής, γιατί η Πολωνία ήταν αυτή που πρώτη άνοιξε τα σύνορά της για να υπάρξει η νέα γερμανική μεταπολίτευση και η πανένωση των Γερμανιών. Και τελικά βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια. Μιλάμε για συνταγματικές παραβιάσεις, για παραβιάσεις του συνταγματικού δικαίου. Μιλάμε για διάφορα εργαλεία, για πάγωμα χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μπορούμε να, να τα κάνουμε. Δεν λέω όχι, αλλά αυτό που βασικά χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος στην χώρα αυτή, διότι αν δεν μιλήσουμε με τους πολίτες της Πολωνίας ή και τους πολίτες των δικών μας χωρών που αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται απλά για μια γραφειοκρατική αιμονή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα. Γι' αυτό και χαραζόμαστε ένα πραγματικό, ειλικρινή διάλογο για το κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα. Πρόεδρος, δύο συντονιστές έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ γρήγορα γιατί υπάρχουν και άλλα τρία μέλη της ε, Επιτροπής μας και έχουμε και άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε και έχουμε υπερβεί το χρόνο. Κυρία Ζήπελ, σας παρακαλώ πολύ, μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, απλώς θέλω να τονίσω αυτό που είπε η συνάδελφος Τέρι Ράιντκε όταν μίλησε για το κράτος δικαίου. Γιατί πράγματι πρέπει κανείς πάντοτε να μιλά πάντοτε για το τρίγωνο. Το κράτος δικαίου προστατεύει τη δημοκρατία και εξασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όμως και τα τρία είναι αλληλένδετα και ανήκουν στο ίδιο σύστημα. Γι' αυτό και ε, θέτουμε αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται και με την ε, απαράδεκτη δημιουργία ζωνών ελεύθερων από ΛΟΑΤΚΙ. Είχαμε στο παρελθόν αντίστοιχα πράγματα για Εβραίου. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει επίση κάποια ε, ΛΟΑΤΚΙ ιδεολογία. Αν ερωτευτείς άντρα ή γυναίκα, τότε αυτό απλώς σου συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο το πιστεύεις, δεν είναι κάποια πεποίθησή σου. Δεν μπορεί κανείς να προσχωρήσει σε μια πεποίθηση ότι αύριο θα ερωτευτεί μια γυναίκα ή έναν Άντρα, Δεν πρόκειται λοιπόν περί ιδεολογίας, πρέπει να σταματήσει αυτή η ρητορική. κυρία Ίντβελτ, σε ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω ότι παρά τι δηλώσει περί του αντιθέτου που ακούμε από του Πολωνούς συναδέλφου, φυσικά και βλέπουμε ότι σκόπιμα η πολωνική κυβέρνηση στραγγαλίζει τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και οποιαδήποτε αντιπολιτευόμενη, αντίθετη με εκείνη φωνή. Σταματήστε λοιπόν αυτό που κάνετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή απάντηση. Ελπίζω η, Επιτροπή να κάνει τέσσερα πράγματα διαφορετικά. Πρώτον, να δρά πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνο είναι χρήμα. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι μη αναστρέψιμα. Δεύτερον, το πλήρε πεδίο του άρθρου 2 πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταδείξει κανείς τις συστημικές παρεμβάσεις του άρθρου 2. Τρίτον, Κοιτάξτε και το ζήτημα της διαφθοράς, γιατί πολλέ πολλές φορές μιλάμε για αξίες και κράτος δικαίου κτλ. Όμω Όμως αυτές οι κυβερνήσεις προσπαθούν να καλύψουν το γεγονός ότι είναι διεφθαρμένες μέχρι το μεδούλι και αξιοποιούν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξαγοράζουν την υποστήριξη. Και τέλος, δεν μπορούμε τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις να τις αναθέτουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν το έχει κάνει επίση σε ένα βαθμό. Ελπίζω να το κάνει και το Συμβούλιο. Η διερμηνία τελειώνει, λέει ο Πρόεδρο, και ξέρετε πώ συνεχίζουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Συνεχίζουμε μόνο στα αγγλικά. Κυρία Στρίκ, ένα λεπτό. The, the, the judge... Ευχαριστώ. Οι αποφάσει ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρε. Το ανώτατο δικαστήριο τη Πολωνία ε, μίλησε ξεκάθαρα αλλά οι δράσει τη ε, πολωνική κυβέρνηση επίση ήταν σαφεί. Δεν πρόκειται να σεβαστούν ε, την ομολογία. Αυτό ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ζητάω από τον κύριο Ρέιντερ να μας πει αν έχει αν θα ζητήσει προσωρινά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να σταματήσει η δράση του πειθαρχικού αυτού σώματος το συντομότερο δυνατόν και να προστατεύσετε την ανεξάρτητη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Επίσης, να σας υπενθυμίσω την ερώτησή μου για τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη και την αρμοδιότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 259 εναντίον της Πολωνίας. Η κυρία Βυσνιέσκα. Τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Η Πολωνία είναι ένα δημοκρατικό κράτος. Με κράτος δικαίου. Και θέλω να τονίσω ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 7 εναντίον της Πολωνίας είναι μια διαδικαστική κατάχρηση, αγαπητέ Επίτροπε, όταν βλέπουμε την κατάσταση επικρατεί σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί το άρθρο 7 δεν έχει ενεργοποιηθεί αντίον της Μάλτας, Φερρυπίν, όπου δολοφονούνται δημοσιογράφοι. Γιατί το άρθρο 7 δεν έχει χρησιμοποιηθεί αντίον της Γαλλίας. Και στη Γαλλία περιστέλλονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών για διαδηλώσεις. Πολλοί πολίτε έχουν ε, τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αυτό που προτείνουμε για να ε, τιμωρούμε τους δικαστές υπάρχει και στη Γαλλία. Ίδιος νόμος είναι. Γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 εναντίον τη Γαλλίας. Ένα λεφτό ο καθένας, έτσι. τώρα, η επόμενη γύρα και μετά οι ομιλητές. Σας ευχαριστώ για τα επιχειρηματά σας, ε, Υπουργέ και Επίτροπε. Θα συνεχίσω στα πολωνικά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η τρέχουσα κατάσταση στην Πολωνία δείχνει ότι οι μηχανισμοί επαλήθευσης δεν είναι επαρκείς. Θα πρέπει να, ζητήσουμε, να διαρωτηθούμε εάν οι εθνικές λύσεις σέβονται το ενωσιακό δίκαιο, τους ενωσιακούς μηχανισμούς. Οι ενωσιακοί μηχανισμοί δυστυχώς είναι πολύ αδύναμοι. Υπάρχουν fake news, υπάρχει α, χειραγώγηση, υπάρχει δημιουργία ψευδών ειδήσεων. Είμαστε συχνά πολύ αργοί και δίνουμε τη δυνατότητα για παρερμηνίες. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι ξεκάθαροι σε όλους τους πολίτες και θα είναι ίδιοι παντού. Εάν διορθώσουμε τις διαδικασίες, θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ε, να καταλάβουν ποια είναι τα συμπεράσματα. Θα πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι αυτές οι περίπλοκες δημοκρατικές καταστάσεις. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Πολωνία είναι υπέρ της α, δημαγωγίας. Είμαι Πολωνίδα δικηγόρος. έχω ασχοληθεί με ανθρώπινα δικαιώματα και μακάρι να μην χρειαζόταν να συζητήσουμε την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά η βελτίωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία δεν λαμβάνει χώρα. Στην πρόσφατη επιστολή ε, αναφέρατε ότι γίνονται διάφορες επιθέσεις εναντίον οργανώσεων και ακαδημαϊκών. Ε, η καταστολή εναντίον των ανεξάρτητων δικαστών και εισαγγελίων έχει δατικοποιηθεί την, τις τελευταίες εβδομάδες. Το νομοσχέδιο για την ε, Πισταρχικές δράσεις εναντίον των δικαστών είναι ένα, μια περαιτέρω περιστολή της ανεξαρτησίας των δικαστών. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν έχει τελειώσει, θα τη ζήσουμε και θα την ξαναζήσουμε, γιατί τα κράτη-μέλη, διάφορα κράτη-μέλη, πιστεύω ότι μπορούν να δράσουν με ατιμορρησία. Κυρία Κέμπα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διερωτώ με. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν τι θα κάνει όταν δουν ότι υπάρχουν δικαστές που διαδηλώνουν μαζί με πολίτες στο, δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να νικήσει, γι' αυτό κατεβαίνει στον δρόμο. Με βάση το γαλλικό νόμο, το άρθρο 10 προβλέπει την απαγόρεση τη συμμετοχή των δικαστών σε διαδηλώσεις. Οι δικαστές δεν μπορούν να δείξουν αρνητική και εχθρική στάση απέναντι στην κυβέρνησή του. Γαλλικός νόμος είναι αυτός. Οι δικαστές δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε πολιτικές συγκεντρώσεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Πολωνία. Οι Πολωνοί δικαστές αμφισβητούν τη, την, τους διορισμούς του, από των διαφόρων δικαστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε και θα ήθελα να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό. Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάποιοι από εμά μπορεί να μην ε, συμμεριζόμαστε ε, τις ε, αρχές αλλά πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε τους ε, Πολωνούς δικαστές ε, που τους καταπιέζουν, που τους δυσφημούν και τους ταπεινώνουν τα μέσα με πραγματικά συκοφαντική με συκοφαντικά δημοσιεύματα τα μέσα και ενημέρωση. Μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν ακριβώ ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά όμω πρέπει αυτή να εφαρμοστεί. Έχει προτείνει το πολωνικό Κοινοβούλιο ένα νόμο που ουσιαστικά δεν θα επιτρέψει στους δικαστές να καταθέτουν προδικαστικά ερωτήματα και αν διαφωνούν με τις αρχές ε, μπορεί και να πάβονται από το αξιωμά τους, ε, από το λειτουργήμά τους. Ε, θα, χρησιμοποιήσουμε, θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχουν κάποιες άλλες δυνατότητες, ασφαλιστικές δικλήσεις κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό σώμα του δικαστηρίου. Θα ζητήσετε ασφαλιστικά μέτρα θα έρθετε να δείτε με τα μάτια σας τι γίνεται στην Πολωνία, πρόεδρος. Παρακαλώ να είστε λογικοί. Είχατε το χρόνο σας και τον υπερβήκατε κιόλα, κύριε Γιάκη. 30 δευτερόλεπτα σας δώσω μόνο. Γιατί θέλουμε να ξαναδώσουμε το λόγο στα μέλη του ε, πάνελ και έχουμε και τη Μάλτα μετά. 30 δευτερόλεπτα. Państwo, czy wiecie, że w Polsce orzeka w tej Στην Πολωνία έχουμε 750 δικαστές που έχουν διοριστεί. Και το αποκολλείται αυτό απολυταρχικό καθεστώς. Στη Γερμανία τι ακριβώς έγινε. Το ξέρετε ότι εξαρθρώθηκε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος σε, σε πολωνικό δικαστήριο. Δύο λεπτά, Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι ο πρώην ηγέτης της ε, αντιπολέτευσης στο Κοινοβούλιο θα έκαναν ό,τι τους έλεγε εκείνος αυτή είναι η αμεροληψία για, αυτή, για, για, την οποία μιλάτε. Πρόεδρος, τρία λεπτά και προφανώς τη Μάλτα θα τη ζητήσουμε μόνο στα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στην κυρία Σκτρικ για το ερώτημα Η διαδικασία του 259 είναι μια διαδικασία που ενεργοποιείται από, το κράτος μέλος, όχι από την Προεδρία. Και συμφωνώ με την κυρία Ζίπελ ότι πρόκειται για ένα τρίπτυχο. Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό από εμένα. Εύχομαι αντοχή και επιτυχία στον κύριο Ρέιντερς στη δουλειά του τα επόμενα πέντε χρόνια ως Επίτροπος. Ευχαριστούμε κυρία Τουρπουλάιν, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Ρέιντερς, ναι, πολύ σύντομα. Τα ενδιάμεσα μέτρα Στην τελευταία διαδικασία επί η Κομισιόν ζήτησε επιταχυμένη διαδικασία. Δεν ε, κρίθηκε επιθυμητό όμως κάτι τέτοιο. Ακούω λοιπόν ότι ζητούνται τώρα, ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Για την έναρξη της διαδικασίας άρθρου 7, η Κομισιόν έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα της δικαιοσύνης. Βεβαίω, το παιδί δεν μα περιορίζει. Μπορούμε να, να συζητήσουμε την έναρξη του άρθρου 7 και σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Και, όπως είπα, στην νέα Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται επί όλων αυτών και θα προσπαθήσουμε να, κάνουμε μια, να φτιάξουμε ένα μηχανισμό χωρίς διακρίσεις εναντίον κανένας κράτους μέλους. Ευχαριστώ πολύ. ήταν σύντομο, κύριε Πιτρόπη. Σα ευχαριστώ. Σα εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όμως. Έχουμε τη Μάλτα. Δυστυχώς εδώ η διερμηνία ολοκληρώνεται. Καλό σας βράδυ από τις διερμηνείς. Yes. Thank you. Welcome. Thank you. Christmas. See you in the plenary. See you, in the See you all tomorrow in the plenary. Commissioner, if you want to stay, if you want to stay, well, if you more than welcome, more than welcome. But let's see, let's see. We've got, we've got